Καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Θα συνεχίσουμε με την συνεδρίαση της Επιτροπής μας και φτάνουμε στο σημείο 7 της ημερήσιας διάταξης. Τον ε, κατάλογο που αφορά τις, ε, τη διαρροή άνθρακα, τη μετεκατάσταση των εκπομπών. χθες το βράδυ έλειπαν αρκετοί ε, και ζητήθηκε από τις ε, ομάδες να γίνει σήμερα η ψηφοφορία ή σήμερα το απόγευμα. Επιθυμία ήταν τέλος πάντων να έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε τον κύριο Δήμα στο θέμα αυτό πριν και πριν διακόψουμε το μεσημέρι, για παράδειγμα 12 ε, και 4 με 12 και 25, να ψηφίσουμε ε, το ψήφισμα. Ο συνάδελφος ε, Ζίβερ θέλει το λόγο. Ναι, κύριε Πρόεδρε, χθε εγκρίναμε την ημερήσια διάταξη όπως μας την μοιράσατε και νομίζω ότι αν μεταφέρουμε μία τόσο... αν μεταφέρουμε τώρα ένα τόσο σημαντικό θέμα, Πιστεύω ότι χρειάζεται μια επίσημη απόφαση, διότι διακυβεύονται πολλά στην ψηφοφορία αυτή. Η πολιτική μου ομάδα μπορεί γενικά να δεχτεί αναβολή της ψηφοφορίας, θα πρέπει όμως να διασφαλιστεί σήμερα στις 12 και 4, 12 στις 12 ή 12 και 4 να γίνει η ψηφοφορία. Δεν μπορούμε να δεχτούμε να αναβληθεί για το απόγευμα ή αύριο. Βέβαια, ω προ την ουσία, πιστεύω ότι έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι ενδιαφέρον να ακούσουμε πρώτα τον Επίτροπο. Θα... Ήθελα όμως επί της αρχής ε, να ε, ε, ενημερώνεται ή να, ε, να συμμετέχουν και οι συντονιστές σε μια τέτοια απόφαση. Ευχαριστώ συνάδελφε Ζήπερ. Συμφωνούμε, δηλαδή δεν θα αναβάλουμε για το απόγευμα ή για αύριο την ψηφοφορία. Θα ψηφίσουμε σήμερα το μεσημέρι πριν διακόψουμε. δεν χρησιμοποίησαμε την διαδικασία των διαδρόμων της διάδοσης. Ε, το βράδυ λάβαμε τη σχετική απόφαση. Οι παρόντες συμφώνησαν να κάνουμε αυτή τη μικρή αναβολή. Ωραία, φτάνουμε λοιπόν ε, στην ε, συζήτηση για το θέμα αυτό. Και θα ήθελα να παρακαλέσω αυτούς που υπέβαλαν το ψήφισμα να πάρουν το λόγο. Και Όποιον άλλον ε, θέλει να μιλήσει, να στείλει το λόγο. Ε, σαν του χάσει. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το συζητήσαμε αυτό ήδη στο παρελθόν και νομίζω ότι έχουν ήδη υποθεί τα σημαντικά στη συζήτηση αυτή. να συνοψίσω τα βασικά προβλήματα της απόφασης αυτής της διαδικασίας της Επιτροπολογίας. Θα ήθελα να θυμίσω στους συναδέλφους το θέμα της ε, κατανομής των ε, αδειών για εκπομπές ε, στη βιομηχανία, των δωρεάν αδειών. Το Κοινοβούλιο Θεωρεί ότι ε, η διαδικασία που θα ακολουθείτε θα πρέπει να είναι η δημοπράτηση. Υπήρχε σαφή πλειοψηφία στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και υπήρχε επίσης σαφή πλειοψηφία στην Επιτροπή βιομηχανία. υπέρ της δημοπράτησης. θα μπορούσαμε να δεχτούμε σύστημα όπου οι τομείς ή υποτομείς που διαπιστωθεί μετά από προσεκτική ανάλυση ότι υπάρχει ότι στους τομείς αυτούς υπάρχει κίνδυνος διαρροής άνθρακα, ε, να λαμβάνουν αυτομάτως άδειες. Η βασικές αποφάσεις στο θέμα αυτό ελήφθησαν ουσιαστικά στην Σύνοδο Κορυφής από τους Πρωθυπουργούς. Δεν ακολουθήθηκε η κανονική νομοθετική διαδικασία. Ο συμβιβασμός που επιτεύθηκε ήταν τα κριτήρια για τη διαρροή άνθρακα να είναι αρκετά Εβραία, ώστε οι περισσότεροι να πληρούν τα κριτήρια αυτά. Ωστόσο, ως κομμάτι της ως κομμάτι του συμβιβασμού αυτού ήταν να λαμβάνονται υπόψη οι δράσεις τρίτων χωρών όταν αξιολογείται η διαρροή άνθρακα και οι δεσμεύσεις τους αλλά και η, αποτελεσματικότητα, η ενεργειακή αποτελεσματικότητα του βιομηχανικού τομέα στις τρίτες χώρες. Αυτό ήταν μία πτυχή του συμβιβασμού που δεν έχει εφαρμοστεί, δεν έχει ενσωματωθεί στον κατάλογο των τομέων όπως τον έχει συντάξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου λέει ότι δεν υπάρχουν σαφείς νομικές βάσεις. Αυτή είναι η δική τους αξιολόγηση. Αυτό όμως το θέμα δεν είναι να ε, προσφύγουμε στα δικαστήρια κατά της Επιτροπής. Το θέμα είναι η εφαρμογή ενός νομοθετήματος που έχει υιοθετηθεί με τη διαδικασία της συναπόφασης σύμφωνα με τους στόχους. Ο κατάλογος των τομέων και επιμέρους τομέων δεν είναι ικανοποιητικός και όπως είπε εκπρόσωπος της Κομισιόν στη συνάντηση όπου συζητήσαμε το θέμα αυτό, θα μπορούσε πιθανότατα να εφαρμοστεί σωστά, ώστε να λαμβάνονται υπόψη δηλαδή οι δράσεις των τρίτων χωρών κατά τον καθορισμό των ποσοστών όσον αφορά τα κριτήρια των διαφόρων τομέων. Και ένα πολιτικό θέμα. Πιθανότατα οι συνάδελφοι που επισκέφτηκαν τι Ηνωμένε Πολιτείε την προηγούμενη εβδομάδα, εγώ δεν ήμουν εκεί, και δεν ξέρω αν αναφέρθηκε αυτό, αλλά μπορεί να προσέξατε και είναι γεγονός ότι στη συζήτηση στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει χρησιμοποιηθεί ως επιχείρημα το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κατανέμει ελεύθερα άδειε και αυτό ήταν επιχείρημα στις Ηνωμένε Πολιτείες από την πλευρά αυτών που θέλουν ε, ε, αποδυναμωμένη περιβαλλοντική νομοθεσία εκεί. Μένουν λίγες εβδομάδες μόλις μέχρι την ε, κλιματική σύνοδο της Κοπεχάγης και θα ήταν ατυχές μήνυμα από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν το Κοινοβούλιο συμφωνήσει σε μια απόφαση που θα σημαίνει ότι το 70% των εκπομπών που καλύπτονται από την ε, οδηγία για την εμπορία εκπομπών να αποτελούν αντικείμενο ε, ελεύθερης αδειοδότησης. Υπάρχουν σαφείς λόγοι γιατί το Κοινοβούλιο θα πρέπει να μπλοκάρει την απόφαση αυτή. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, ο κατάλογος θα χρειαστεί την 1η Ιανουαρίου, θα μας χρειαστεί την 1η Ιανουαρίου του 2013. Υπάρχει λοιπόν αρκετός χρόνος να ανασυνταχθεί ο κατάλογος ώστε να ληφθούν υπόψη όλα τα κριτήρια που συμπεριλαμβάνονται στην νομοθεσία. και υπάρχει επίση αρκετός χρόνος ώστε να διασφαλίσουμε ότι ο τελικός οριστικός κατάλογος τη 1 η Ιανουαρίου του 2013 θα λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα των διεθνών διαπραγματεύσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Σατουχάση. Είπατε για γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας για το θέμα αυτό, αλλά τελικά δεν είναι μόνο νομικό, είναι και πολιτικό έτσι, το ζήτημα το πώς θα αντιδράσουμε. Σε ό,τι αφορά τις Ηνωμένε Πολιτείες, αύριο το πρωί θα το ξανασυζητήσουμε. Ο νόμος Πόξα Κέρι προβλέπει ε, δασμούς άλλο ε, μέσο. Αυτό δείχνει ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, έχουν και άλλα μέσα τα οποία μετέρχονται για να προστατεύσουν την ίδια τους βιομηχανία. Αλλά δεν γίνεται με τέτοια μέτρα να έχουμε νομοθεσία για το κλίμα. Ξέρω εγώ και αυτό το border tariff να γίνει climate tariff, δεν ξέρω. Ο Καρλ Χάιντς Φλόρενς πρώτος και έχουμε και άλλους μετά συναδέλφους. Ευχαριστώ. Εκτιμώ πάρα πολύ την κυρία ε, Σάτου Χάτσι, αλλά θα ήθελα να την παρακαλέσω πάρα πολύ όταν μιλάμε για την πολιτική βούληση την περασμένη θητεία να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Διότι η πολιτική βούληση εδώ στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ήταν σαφής και έλεγε ότι θα πρέπει να κάνουμε ένα κατάλογο με θέμα τη διαρροή ε, ε, τη λεγόμενη του διοξιδίου των άνθρακα, carbon Linkage, όχι τέλος του 2009, το λέει το κείμενο αυτό. Και εμείς είπαμε ότι επειδή γνωρίζουμε ότι πρέπει να προχωρήσει η Ευρώπη, θέλουμε βεβαίως να δώσουμε πιστοποιητικά. Όλο το σύστημα των οροφών και των ορίων των ΚΑΠ παραμένει. Απλώς αναβάλλεται ο πληστηριασμός για τις άδειε μέχρι να δούμε πώς θα αντιδράσουν ε, οι ε, άλλες μεγάλοι ε, ήπειροι στη γη μας. Δεν είναι σωστό λοιπόν να λέμε ότι δεν υπήρχε πολιτική βούληση. Το ETS, το σύστημα εκπομπής, ε, δεν θα είχε ποτέ ε, γεννηθεί εάν δεν το είχαμε συνδέσει ακριβώς με τις βιομηχανίες που φεύγουν επειδή ρηπαίνουν. Και ε, ανεξάρτητα με το μήκος του καταλόγου, δεν μπορώ να το κρίνω, πάντα Εκπλήσουμε πάρα πολύ που μπορούν να το κάνουν άλλοι συνάδελφοι. Εγώ προσωπικά δυνατό. Επαφίεμαι στη ε, πραγματογνωμοσύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχει πολλούς εμπειρογνώμονες και συλλέγει πολλά στοιχεία. Εκεί λοιπόν βασίζομαι εγώ και προσανατολίζομαι και πιστεύω ότι πρέπει η μέρα να εγκρίνουμε τον κατάλογο. Α, να πω και δύο λόγια για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ακριβώς οι Αμερικανοί ήξεραν ότι εμείς δεν ε, προτιμούμε αυτό το θέμα των δασμών στα σύνορα, αλλά ε, το ETS. Σε αντίθεση με τα όσα είπε η κυρία Χάση, όσο δεν υπάρχουν ε, διεθνείς ρυθμίσεις και αξιόπιστη σύμβαση, προτιμούμε να αναβάλουμε αυτή τη δημοπρασία, τον πληστηριασμό. Εγώ νομομαθής δεν είμαι, αλλά έχω και στην πολιτική μου ομάδα και στο φίλο μου νομομαθείς που μου εξηγούν το κείμενο και μου το ερμηνεύουν και καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει λόγος να καταψηφίσει κανείς αυτή την πρόταση για την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ δεν θέλω να καταρρύψω αυτό το έγγραφο ε, με νομικά επιχειρήματα. Υπάρχουν αρκετά πολιτικά επιχειρήματα για να το κάνει κανείς αυτό, αλλά θα αρκούσαν και μόνο τα νομικά για να καταπέσει ε, και να το ε, απορρίψουμε. Λοιπόν, εμείς είμαστε ακριβώς στο πνεύμα της συζήτησης που είχαμε κάνει για τα δικαιώματα εκπομπής ρήπων και το εμπόριο. Αυτό το συζήτησε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τήρησε το λόγο της. Τώρα δεν ξέρω αν τήρησε παντού το λόγο της. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Για το συγκεκριμένο όμως είμαι πολύ υπέρ του να καταψηφιστεί το ψήφισμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ ο Κρίς Ντέβις. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε ο κατάλογος που πρέπει να εξαιρεθεί από τον πληστηριασμό είναι τόσο μεγάλος που στην ουσία ε, ε, υποσκάπτει ολόκληρη την αρχή. Αλλά από τη στιγμή που είναι ο στόχος να επιτύχουμε 25% μείωση στο διοξείδιο του άνθρακα, ε, δεν είμαι βέβαιος πως έχει νόημα αυτό, γιατί αυτό είναι πολύ εύκολο να επιτευχθεί. Το ίμιση του 25% μπορεί να επιτευχθεί αγοράζοντας πιστώσεις απαλού. Ένας στόχος τόσο λίγο φιλόδοξος μπορεί απλά να επιτευχθεί μέσω της χρήσης ε, του EST, ε, ETS μάλλον, μέσω της εξοικονόμησης απλής ενέργειας. Ε, είναι πραγματικά ελάχιστα φιλόδοξο αυτό το πρόγραμμα. Είτε το υπερψηφίσουμε ή το καταψηφίσουμε αυτό το ψήφισμα δεν έχει και πολύ νόημα, γιατί αφού μιλάμε μόνο για 20% μείωση είναι αποτυχία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση από μόνη της δεν μπορεί να σώσει τον κόσμο από τις κλιματικές αλλαγές. Πρέπει να υπάρξει διεθνή συμφωνία και πιο φιλόδοξη από ό,τι είχαμε μέχρι στιγμής. Και αν θέλουμε να γίνει η διεθνή συμφωνία, να υπάρξει η διεθνή συμφωνία, τότε θα πρέπει να ξέρουμε πως ο δικός μας ο στόχος θα πρέπει να αυξηθεί από το 25% στο 40%. Οπότε η Κομισιόν θα πρέπει να επανέλθει με νέες προτάσεις και θα ε, ε, χρειαστεί να αναγνωρίσει πως η βιομηχανία θα πρέπει και αυτή να πληρώσει κάποιες συνέπειες για την μεγαλύτερη, και η μεγαλύτερη χρήση του πληστηριασμού είναι από τους τρόπους ώστε να διασφαλίσουμε πως ισχύουν σωστά οι αρχές του ETS. Το πραγματικό πρόβλημα είναι πότε θα γνωρίζουμε αν η Κομισιόν θα επανέλθει με κάποιο πιο ε, χτενισμένο κατάλογο και αν θα έχουμε input. Θα έχουμε... Εμείς δεν, δεν συμβάλαμε στην προετοιμασία αυτού του καταλόγου. Εμείς ε, προετοιμάσαμε το πακέτο για την κλίμα. Η Λίντα Εύα ήταν κομμάτι της ε, διαπραγματευτικής ομάδας και τελικά το πακέτο πήγε στους υπουργούς, πήγε στο Συμβούλιο. Δεν είχαμε ευκαιρία να το τροποποιήσουμε μετά. Απλώς ψηφίσαμε για το πακέτο των κλιματικών αλλαγών unblock. Ολόκληρη διαδικασία συναπόφασης τελικά που έπρεπε να έχει γίνει, ε, είχαμε, ε, έγινε με ελάχιστη συμβολή από την Επιτροπή μας. Άρα λοιπόν θα πρέπει να γίνει τώρα. Αν πετύχουμε συμφωνία στην Κοπεχάγη σε κάποια επόμενη διάσκεψη τον επόμενο χρόνο, τι θα κάνει η Κομισιόν. Νομοθεσία δεν είναι ξεκάθαρη. Το θέμα είναι πότε θα υποχρεώσουμε την Κομισιόν να επανέλθει και να κάνει νέε προτάσει. Εγώ να κάνω προτάσει. Εμεί κάνουμε κάποιε χειρονομίε. Από τη στιγμή που μιλάμε μόνο για 20% μείωση στην, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι απλά ένα διαπραγματευτικό χαρτί, είναι μια χειρονομία για να βοηθήσουμε στην επίτευξη μια διεθνού συμφωνία. Εγώ θέλω να ξέρω, θέλω συγκεκριμένη δέσμευση από την Κομισιόν ότι θα επανέλθει, θα παρουσιάσει νέε προτάσει πιο φιλόδοξε και σε κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Αν δεν το πάρουμε αυτό, ε, τότε θα είμαστε κατά του ψηφίσματο. Αν ο Επίτροπο Δήμα μπορεί να μα δώσει τέτοιου είδου εγγυήσει όταν θα μιλήσει αργότερα, τότε εντάξει. Αν όμω όχι, τότε θα κάνω τη δική μου χειρονομία σήμερα και θα υπερψηφίσω το ψήφισμα αυτό και θα θυμίσω απλά στην Κομισιόν και στο Συμβούλιο πώ θέλουμε να ε, μας λαμβάνουν υπόψη και θέλουμε συγκεκριμένες δεσμεύσεις για το ότι οι φιλοδοξίες που γενικόλογα εμείς έχουμε δεχτεί και υποστηρίζουμε θα πρέπει να ισχύουν και για τις λεπτομέρειες. Η Λίντα Μακέβαν. Καταρχήν θέλω να πω ότι δεν πρέπει να αρχίσουμε να κάνουμε, να μιλάμε μάλλον για θεωρίες συνωμοσίας. Δεν είναι αλήθεια πως δεν συμμετείχαμε στην νομοθεσία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας των Εκπομπών. Όχι. Δεν είναι αλήθεια. Η γιατί ήμουν εκεί, ήμουν εκεί στους τριμερείς διαλόγους, συζητήσαμε εδώ στην Επιτροπή, το ψηφίσαμε τον Οκτώβριο, έπειτα εβδομάδες επί εβδομάδα ε, γίνονταν τριμερείς επαφές και στην ομάδα μου είχαμε ατελείωτες συζητήσεις για όλες τις λεπτομέρειες. Ποτέ δεν έχουμε συζητήσει κάτι τόσο πολύ όσο το ETS στο Κοινοβούλιο. Και όλες τις λεπτομέρειες συζητήσαμε. Ας μην λέμε πως αυτά όλα τα φτιάξαν οι, προ... οι πρωθυπουργοί. Ε, ε, αρχικά αυτή η επιτροπή, την ημέρα που ψήφισε αυτή η επιτροπή, αν θυμάμαι καλά, ήταν, ήταν Ιούνιος 2010 και αυτό έχει νόημα γιατί ακριβώς τότε αρχίζει να ισχύει και το άρθρο 10β που λέει ότι η Κομισιόν υπό το φως των διεθνών διαπραγματεύσεων θα παρουσιάσει ένα κατάλογο τομέων ε, κλάδων μαζί με τους τομείς του, της Διεθνούς Συμφωνίας. Αυτό έχει νόημα. Αλλά είναι και τμήμα της πολιτική ε, συμφωνία εδώ που προχωρήσαμε στο Μάρτιο του 2010. Ήδη δηλαδή η Επιτροπή Περιβάλλοντος κατάφερε να φέρει πιο μπροστά την ημερομηνία. Μάρτιο 2010 και έπειτα στι συζητήσει του Συμβουλίου, όχι στη διάσκεψη κορυφή του Συμβουλίου, το Δεκέμβριο του 2009 και πολλοί κόσμος από τον κλάδο τους πίεσε ε, και έχουν μάθει πλέον ότι το να πιέζουν για αυθαίρετες ημερομηνίε δεν είναι πολύ σοφό. Γιατί μετά βλέπουμε τι αποτελέσματα δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα να φτιαχτεί αυτό ο κατάλογο μέχρι το τέλο του χρόνου. Και από εκεί προήλθε αυτή η ημερομηνία και αποφασίστηκε στου τριμερεί διαλόγου, όχι στην διάσκεψη ε, στο Συμβούλιο Κορυφή. Εκεί αποφασίστηκαν ε, τρία-τέσσερα θέματα, αν θυμάμαι καλά. Το ένα ήταν ουσιαστικό, ότι δηλαδή οι δωρεάν ε, ποσότητε για άδειε θα δίνονταν ανάλογα με τον ε, με τις επιχειρήσεις. Αυτό, δεν, αυτό ήταν ένα από τα πιο ουσιαστικά. Τα υπόλοιπα δεν ήταν τόσο σημαντικά, αλλά μην λέμε ότι δεν αποφασίστηκε δημοκρατικά η νομοθεσία αυτά. Η δική μου ομάδα, ωστόσο, είναι διχασμένη για αυτό το θέμα και θα ακούσουμε πολύ προσεκτικά τα όσα θα μα πούν οι εκπρόσωποι τη Επιτροπή σήμερα και τα όσα θα μα πει και ο κύριο ε, Δήμα, ο Επίτροπο. Θα ήταν ωραίο να δούμε μόνο την πολιτική πτυχή του συστήματος αυτού, γιατί εγώ μπορώ να πω ότι ποτέ δεν ήθελα τον Ιούνιο, ποτέ δεν ήθελα τον Δεκέμβριο και πιστεύω πως αυτός ο κατάλογος είναι εξαιρετικά μακροσκελής. Αλλά αυτό είναι θέμα επιτροπολογίας, δεν είναι πολιτικό ζήτημα αυστηρά και αν πούμε όχι σήμερα, αν τον απορρίψουμε τον κατάλογο σήμερα θα πρέπει να πάμε στην Ολομέλεια και αν πάμε στην Ολομέλεια και απορρίψουμε πάλι τον κατάλογο τότε ανοίγουμε νομικές ερμηνείες για αυτό που κάναμε. Πρέπει να αναλύσουμε την νομιμότητα των όσων κάναμε σύμφωνα με την την νομοθεσία που έχουμε υιοθετήσει. Είμαστε κοινοβούλιο εδώ πέρα μέσα και πρέπει να τηρούμε την νομοθεσία. Αυτό που χρειαζόμαστε λοιπόν σήμερα το πρωί από την Κομισιόν είναι η σαφήνεια για το γιατί δεν έλαβαν υπόψη τις πληροφορίες της χώρας. Τι πληροφορίες ζήτησαν, είναι αυτά που έχει στο 10α της νομοθεσίας. Μετά, πώς θα λειτουργήσει το 10β, το άρθρο 10β που ξέρουμε ότι έχει αναφερθεί στα... και από τα λόμπι είναι ένα πολύ σημαντικό άρθρο μέσα σε αυτή την νομοθεσία. Λέει ότι η Κομισιόν μέχρι τον Ιούνιο φέτος θα πρέπει μέσω διεθνού συμφωνίας να ορίσει το τμήμα των αδειών που δίνεται δωρεάν στους τομείς και ποιους υποτομείς, σε ποιους κλάδους ε, θα λειτουργήσει υπό το άρθρο 10α. Πώς το βλέπει η Κομισιόν, ποια μεθοδολογία θα χρησιμοποιήσει για να συστήσει αυτό τον κατάλογο, ε, να συντάξει αυτό τον κατάλογο. Ε, είναι τροπολογία. Εγώ δεν είμαι βέβαιος ότι θέλω να μπω σε όλες τις λεπτομέρειες τεχνικές. Τα δώσαμε στην επιτροπολογία και πρέπει να τη δεχτούμε. Δεν μπορούμε τώρα να αρχίσουμε να λέμε πως ε, να, ζητάμε μάλλον πολιτικό κατάλογο. Θα είναι και μακρύτερος μάλλον και όχι συντομότερος. Τι σημαίνει τώρα το 10α. Μπορεί ο κατάλογος να γίνει μακρύτερος ή, ή μικρότερος. Λέει στην νομοθεσία ότι οι τομεί μπορεί να προσθεθούν στον κατάλογο όταν ε, θα έχει αυτό ε, πια καθοριστεί. Αλλά σε ποια φάση νομικά θεωρείται εγκεκριμένο αυτό ο κατάλογο, τώρα ή μετά την κοπεγάγη. Δηλαδή, ο κατάλογο μπορεί να. Μάλλον μπορεί κάποιο τομέα να αφαιρεθεί από τον κατάλογο μετά από την υιοθέτηση τη Διεθνού Συμφωνία. Και ξέρω πω οι συνάδελφοι θα έχουν και άλλε ερωτήσει για την Κομισιόν. Ε, και η τελευταία μου παρατήρηση είναι ότι δεν πρέπει να τρέφουμε πάτες, ότι αν θέλουμε να δώσουμε δωρεάν άδειε. Αυτό σημαίνει ότι οι βιομηχανίες θα ανασάνουν, αλλά δεν, δεν υπάρχει κάποιο κατόφλι που να μειωθεί. Δηλαδή, ο αριθμός των δωρεάν αδειών θα μειωθεί για όλους τους τομείς που, δίνουν, που μπορούν να έχουν δωρεάν άδειε. Θα υπάρχει δηλαδή και μια σύγκριση μεταξύ των τομέων και μόνο οι πιο αποδοτικοί θα παίρνουν τις δωρεάν άδειε. Και όσοι το ξεπερνούν τα κατόφλια, ούτως ή άλλως θα πρέπει να, πάρουν τα, να, να αναγοράσουν τις αδειε Θα πρέπει η Κομισιόν να μας εξηγήσει. Ε, κάποιος το ρώτησε χθε το βράδυ γιατί είναι το κρασί στον κατάλογο. το κρασί, τι κάνει ο κλάδος, τι εκπομπές έχει ο κλάδος αυτός. Ε, Μιλάμε λοιπόν και επαναλαμβάνω για διαδικασία επιτροπολογίας και ας μην βάλουμε τρικλοποδιά στις διαπραγματεύσεις αυτές. Äh, Ευχαριστώ πολύ, ο Ρίχαρτ Τσίπερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συμφωνήσω με τις ερωτήσεις της Λίντα Εύανς, ειδικά όσον αφορά το άρθρο 10. είναι πολύ περιορισμένα τα δικαιώματα και τα προνόμια του Κοινοβουλίου στον ε, τομέα αυτό, στη διαδικασία της επιτροπολογίας ε, δηλαδή και νομίζω ότι η γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας ε, δείχνει ότι δεν υπάρχουν οι σωστές νομικές βάσεις. Δηλαδή είναι πολύ σαφή τα επιχειρήματα σχετικά με τη μορφή αυτού αυτής της απόφασης. Ο Κάρχανς Φλόρανς πολύ σωστά ε, ερμήνευσε την κατάσταση. Είμαι δηλαδή ε, ως προς τη μορφή κατά της, ε, του ψηφίσματος αυτού. Θα ήθελα όμως επί της ουσίας να σας θυμίσω ότι ε, η βιομηχανία είναι εταίρη μας και κάποιες ε, διαδικασίες αρκετέ διαδικασίε ε, στη βιομηχανία μπορούν να λάβουν πιο αποτελεσματική μορφή και δεν. Είναι σωστό ότι μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει το σύστημα εμπορίας, ούτε καν με τον κατάλογο αυτό. Ε, μόνο το 10% δεν χρειάζεται να αγοράσει επιπλέον δικαιώματα εκπομπών. Η ελεύθερη κατανομή δηλαδή αφορά μόνο το, 10, το καλύτερο 10%. Και η βιομηχανία με την υιοθέτηση του καταλόγου θα πρέπει να γίνει πιο αποτελεσματική να εφαρμόσει δηλαδή πιο αποτελεσματικές διαδικασίες. Η Ευρώπη αντιπροσωπεύει το 10% των εκπομπών παγκοσμίω. Υπό το φως των υποχρεώσεων που έχουμε αναλάβει στην Κοπεχάγη, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι με τον κατάλογο αν δεν υιοθετήσουμε τον κατάλογο αυτό δεν θα κάνουμε κάτι καλό ούτε για το... Δεν θα κάνουμε τίποτα καλό ούτε, ούτε για το κλίμα, ούτε για τις θέσεις απασχόλησης, ούτε για το περιβάλλον, ούτε για την Ευρώπη. Η Κομισιόν νομίζω ότι πολύ σωστά πρότεινε τον κατάλογο αυτό. Ομόφωνα υιοθετήθηκε στο Συμβούλιο Υπουργών θα πρέπει λοιπόν πιστεύω να σκεφτόμαστε αν είμαστε εμείς ε, ο κατάλληλος φορέας να απορρίψει μια τέτοια απόφαση. Εμείς λοιπόν θα καταψηφίσουμε το ψήφισμα, θα, θα ε, ψηφίσουμε υπέρ του καταλόγου. Ευχαριστώ, έχω αρκετούς στον ε, κατάλογο. Ε, συγγνώμη, βλέπω αρκετού ορθίου εδώ πέρα. Έχουμε ζητήσει μεγαλύτερη αίθουσα. Φυσικά υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για μια τέτοια συζήτηση. Επειδή θα ψηφίσουμε, παρακαλώ φροντίστε να έχετε την κάρτα ψηφοφοριών σας. Ευχαριστώ πολύ. Μάρτιν Κάλαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι όσο γίνεται πιο σύντομος. Είναι αρκετά απλό το θέμα. Είτε μας αρέσει είτε όχι. Καταλήξαμε σε μια πολιτική συμφωνία. Συμμετείχαμε στις συζητήσεις στην προηγούμενη θητεία του Κοινοβουλίου. Ε, ως αποτέλεσμα η Κομισιόν ε, μέχρι το τέλος του 2009 υπέβαλε τον ε, κατάλογο των τομέων αυτών. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν ποιο είναι το επιχείρημα αυτών που προτείνουν το ψήφισμα αυτό. Αν λένε ότι δεν συμφωνούμε με τον κατάλογο των, της Κομισιόν, ας ακούσουμε ποιου ποιους τομείς θα ήθελαν να αποκλείσουν από τον κατάλογο αυτό. Η Λίντα ανέφερε τον τομέα του Ίνου. Υπάρχουν όμως και πολλοί άλλοι πολύ σημαντικοί ευρωπαϊκοί τομείς και όλοι θα θυμάστε τη μεγάλη συζήτηση που είχαμε για τη διαρροή άνθρακα. Δεν έχει κανένα νόημα να μετακατασταθούν επιχειρήσεις από την Ευρώπη σε άλλα μέρη του κόσμου και τελικά να καταλήξουμε σε περισσότερες εκπομπές από ό,τι στην Ευρώπη. Και έτσι το μόνο που πετυχαίνουμε είναι να εξάγουμε ένα σωρό θέσεις απασχόλησης. Κατά τη γνώμη μου, λοιπόν, δεν έχει νόημα να απορρίψουμε τον κατάλογο, αν αυτοί που ε, θέλουν να καταψηφίσουμε τον κατάλογο θέλουν να μας προτείνουν ποιοι τομείς θα πρέπει να αποκλειστούν, να το εξετάσουμε αυτό. Μπορούμε επίσης να εξετάσουμε την όλη διαδικασία της επιτροπολογίας, αλλά ζητήσαμε από την Κομισιόν να υποβάλει ένα κατάλογο. Τον υπέβαλε, συντάχθηκε από την Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων, ε, και συμφωνώ με τον Ιχαρτ Σίπερ ότι δεν χρειάζεται να καθυστερήσουμε περισσότερο την κατάσταση. Πολλές επιχειρήσεις ε, περιμένουν να λάβουν αποφάσει σχετικά με το αν θα πρέπει να αυξήσουν την παραγωγή, να μεταφέρουν την παραγωγή, να μειώσουν την παραγωγή. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί όσον αφορά την υιοθέτηση νομοθεσίας που θα τους δώσει κίνητρα να ε, φύγουν από την Ευρώπη. Αυτό δεν συμφέρει κανέναν. Ελπίζω Μπορούμε να ξαναεξετάσουμε το θέμα υπό το φως της Κοπεχάγης, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να υπερψηφίσουμε τον κατάλογο και εγώ θα καταψηφίσω το ψήφισμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Chairman. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι απλό το θέμα. Δεν θέλω να ξαναγράψω την ιστορία. Δεν θέλω να προσθέσω μη στον κατάλογο ή να του αφαιρέσω. Δεν είναι αυτή η δουλειά μου. Η δουλειά μου αυτή τη στιγμή είναι να εξετάσω σε τι βαθμό η Επιτροπή έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει σύμφωνα με την οδηγία που υιοθετήσαμε πέρσι. Δεν με ενδιαφέρει η συζήτηση για το ποιο υιοθέτησε τι. Εγώ είμαι νέο εδώ, διαβάζω την οδηγία που υπάρχει και θα κρίνω τώρα εάν η Επιτροπή έκανε σωστά τη δουλειά της. Και είναι απλή η δουλειά αυτή πρέπει να είναι σαφές ότι εδώ δεν είμαστε απλά νομική υπηρεσία, πρέπει να λάβουμε και πολιτική απόφαση σχετικά με το αν η Επιτροπή έκανε τη δουλειά της. Συμφωνώ με την Λίδα Μακέβαν ότι από τη μία πρέπει να γνωρίζουμε τι λέει η νομική υπηρεσία, από την άλλη όμως θα πρέπει να αναλάβουμε και εμείς τις υποχρεώσεις μας ε, και να κρίνουμε πολιτικά. Και έτσι η δική μου απόφαση είναι απλή και υποστηρίζεται από την νομική υπηρεσία, διότι η νομική υπηρεσία λέει ότι δεν μπορεί να κρίνει σε τι βαθμό είναι σωστό να μην ληφθούν υπόψη οι δράσεις και η αποτελεσματικότητα των τρίτων χωρών. Αναγνωρίζουν ότι αυτά δεν λαμβάνονται υπόψη από την ε, Κομισιόν, συμφωνούν ότι αυτά μπορεί να επηρεάσουν τον κατάλογο και συμφωνούν ότι επιστημονικά δεν μπορούν να κρίνουν αν είναι σωστή απόφαση ή όχι. Είναι πολιτική απόφαση της Επιτροπής μας ε, ε, ε, πολιτική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να υποβάλει τον κατάλογο αυτό μέχρι τα τέλη του 2009, αλλά η, η απόφαση αυτή δεν λέει ότι θα πρέπει να περιλαμβάνει όλε τι επιχειρήσει, λέει ότι θα πρέπει να είναι ένα πρώτο κατάλογο. Κάθε χρόνο μπορούν να συμπεριλαμβάνονται νέοι τομεί, μπορεί κάθε χρόνο να μεγαλώνει ο κατάλογο. Μία πιθανότητα υπάρχει μόνο να μειωθεί ο κατάλογος και αυτή είναι η αξιολόγηση μετά την Κοπεχάγη. Στη συζήτηση που είχαμε στην Επιτροπή μας πριν από μία πριν από ένα μήνα και ρωτήσαμε με ποια κριτήρια θα γίνει η αξιολόγηση, η Κομισιόν είπε δεν μπορούσε να δώσει ε, σαφή απάντηση, είπε ότι δεν ξέρουμε ακόμα. Θα γίνει η αξιολόγηση. Αυτό, αυτή είναι η μόνη δυνατότητα να μικρύνει ο κατάλογος. Ε, επέλεξε λοιπόν πολιτικά η Επιτροπή να κάνει ένα μακρύ κατάλογο αυτή τη στιγμή, επέλεξε να μην λάβει υπόψη τα στοιχεία τρίτων χωρών. Αυτή λοιπόν είναι πολιτική απόφαση και τώρα εναπόκειται σε εμά πολιτικά να αποφασίσουμε εάν έχουμε αντίρρηση στις στι πολιτικέ αυτέ αποφάσει. Και εγώ έχω αντίρρηση στι πολιτικέ αυτέ αποφάσει, διότι πιστεύω ότι στον κατάλογο θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται μόνο οι τομεί και οι επιχειρήσει για τι οποίε γνωρίζουμε σίγουρα ότι θα αποτελούν ε, μέρο ε, τη διαρροή του άνθρακα. Και μετά την Κοπεχάγη ε, θα έχουμε τη δυνατότητα να προσθέσουμε και άλλε επιχειρήσει στον κατάλογο. Πιστεύω λοιπόν ότι λαμβάνονται πολιτικές αποφάσεις εντό τη Επιτροπής με τις οποίες δεν συμφωνώ, διότι δεν ευθυγραμμίζονται με την οδηγία που λέει ότι η πρώτη βάση θα πρέπει να είναι η δημοκρατήση. Αυτή λοιπόν είναι η πολιτική απόφαση που λαμβάνω εγώ εδώ πέρα ως ευρωβουλευτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ε Ρώση. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ ευχαριστώ σε μεγάλο βαθμό με τις παρεμβάσεις των συναδέλφων που προηγήθηκαν, Κάλαναν και σύμπερ. Εγώ θεωρώ πως το να εγκρίνουμε αυτό το ψήφισμα και άρα να αμφισβητήσουμε τον κατάλογο της Κομισιόν θα οδηγούσε σε περαιτέρω απώλεια θέσεων εργασίας για τις ε, Ευρωπαίους πολίτες γιατί οι εταιρείε μας θα μπορούσαν να μετεγκατασταθούν σε άλλες χώρες, χώρες όπου σε αντίθεση με αυτό που υποχρεώνουμε τις Ιταλικές και τις Ευρωπαϊκές εταιρείε να κάνουν δεν σέβονται τους κανόνες καλή συμπεριφοράς για τις εκπομπές. Εγώ πιστεύω πώς έχουν αυξηθεί οι εκπομπές σε τρίτες χώρες όπως η Κίνα για να σας δώσω ένα παραδειγματάκι ε, ενώ περιορίζονται στην Ευρώπη. Και πραγματικά θεωρώ πως αίτιο της μετεγκατάστασης μεγάλων εταιριών είναι αυτή. Άλλοι θεωρούν πως υπάρχουν άλλοι λόγοι. Γι' αυτό πάντως δεν έχει μεγάλη σημασία. Πάντως στην Ευρώπη γίνονται λιγότερες εκπομπές, ενώ σε άλλες χώρες εκπομπέμπουν περισσότερο οι ανταγωνιστές μας δηλαδή. Αυτό το ψήφισμα μπορεί να βλάψει ακόμη περισσότερο τη δικιά μας επικράτεια. Όχι να δώσει μόνο ωφέλη κλιματικά, αλλά να οδηγήσει σε απώλεια θέσεων απασχόλησης. Αυτή το ψήφισμα σε μεγάλο βαθμό παρουσιάζεται από ευρωβουλευτές ε, που ανήκουν σε εκείνο το, το, κομμάτι που το οποίο ανήκει στην αριστερά και που θα έπρεπε να είναι πιο κοντά στις ανάγκες των εργαζομένων της Ευρώπης σε μια τέτοια περίοδο κρίσης. Και άκουσα τους συναδέλφους να λένε ότι α, το πνεύμα της προηγούμενης θητείας όταν ονομοθετήσαμε προς αυτή την κατεύθυνση ήταν ότι έπρεπε να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ναι, αλλά στην προηγούμενη θητεία, αγαπητοί συνάδελφοι, η δεν ήταν αυτό που είναι σήμερα. Τόσε θέσει απασχόληση που έχουν χαθεί ε, σήμερα δεν τι χάσαμε στην προηγούμενη θητεία. Το να συνεχίζουμε και να επιμένουμε σε μια γραμμή που έχει προκαλέσει προβλήματα είναι λάθος. Εμείς σήμερα έπρεπε να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τις εταιρείε μας, όχι για να φύγουν, αλλά για να μείνουν στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια και να δώσουν δουλειά εδώ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν ε, κανείς δεν είναι αντίθετος ότι ναι πρέπει να κάνουμε κάτι για το κλίμα, αλλά όχι στις πλάτες των εργαζόμενων. Άρα λοιπόν ως αντιπροσωπεία της Lega Nord εγώ ε, είμαι απολύτως αντίθετος σε, σε αυτό το ψήφισμα. Θεωρούμε πως ο κατάλογος αυτός μπορεί να βελτιωθεί και να εφαρμοστεί, αλλά ότι δεν μπορεί να ακυρωθεί όπως το ζητά αυτό το ψήφισμα. Ευχαριστώ. Κύριε Ρώση, εχθές ήδη είπα ότι οι θέσεις εργασία σε αυτόν τον καιρό δεν απειλούνται από το κλίμα, αλλά από τη σπέκουλα, την κερδοσκοπία των τραπεζών και των χρηματιστηρίων. Και για τη λίστα μιλάμε για το 2013, που ελπίζουμε μέχρι τότε να έχει ανακάμψει η οικονομία. Οπότε ας μην μπερδεύουμε πράγματα και συγκρίνουμε ανώμια μεταξύ τους. Η κυρία Μπάρμπαρα Ντεμπρούν, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να επανέλθω σε ε, αρκετά μικρά σημεία. Πρώτον, κάναμε πλήρη συζήτηση και εκτενή στην προηγούμενη θητεία. Δεύτερον, εγκρίναμε το πακέτο. Κανείς δεν ήταν πλήρω ικανοποιημένο, αλλά συμφώνησαν όλοι ότι υπάρχει αυτή η δέσμη επιτέλους και ως ε, ενεχόμενο μέρος και ένα τμήμα ήταν να έρθει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας φέρει λίστα μέχρι το Δεκέμβριο του 2009. Κανείς δεν προσπαθεί να ανοίξει ξανά τη συζήτηση με το ψήφισμα. Αλλά όπω είχε καθήκον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να φέρει τον κατάλογο μέχρι τα τέλη του έτου, είχε και καθήκον ο κατάλογος αυτός να βασίζεται σε κάποια κριτήρια. Και εμείς ως, Κοινοβούλιο έχουμε εξίσου ευθύνη να κοιτάξουμε και να μελετήσουμε το εάν και κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο πλήρωσαν αυτά τα κριτήρια και πραγματικά έχουν κάνει σωστά τη λίστα. Έχουν καταρτήσει τον κατάλογο Πάντω είναι γεγονός ότι όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν και να ολοκληρωθούν ε, σύμφωνα με την νομοθεσία. Εμείς κοιτάξαμε τη μα είπε Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, στην πορεία και είναι σαφές πιστεύω ότι ορισμένα κριτήρια δεν έχουν πληρωθεί. Δεν έχει ληφθεί υπόψη ας πούμε, η αποτελεσματικότητα των εργοστασίων σε τρίτες χώρες και των δεσμεύσεων σε τρίτες χώρες και αν δεν έχει εκπληρωθεί αυτό το κριτήριο που κατά την άποψή μας δεν έχει, είναι καθήκον μας ε, ως κοινοβούλιο να τα κατονομάζουμε όλα αυτά. Και είμαστε και εμείς ενεχόμενο μέρος και θα πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι για να προχωρήσει το θέμα αυτό. Λοιπόν, παρακαλούμε, καταρτήστε και πάλι ένα κατάλογο που να πληρεί όμως όλα τα κριτήρια της νομοθεσίας που εμείς έχουμε θεσπίσει. Ευχαριστώ, κύριε Λίζε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και πάλι να υπογραμμίσω αυτά που είπαν οι Φλόρεντς και Ζέμπερ και να σας εμ, διευκρινίσω κάποια επιχειρήματα. Ακόμα και αν δεν είναι αποφασιστικό αυτό, θα πρέπει να ξέρουμε τι έγινε πέρσι στην νομοθεσία. Είπε η του και σωστά, ότι και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και στην Επιτροπή Βιομηχανίας είχαμε διαφορετική ψηφοφορία και διαφορετικό αποτέλεσμα για το carbon leakage από αυτό που έχουμε σήμερα. Το θέμα όμως δεν, σημαίνει αυτό, ούτε πρέπει κανείς να συμπεράνει ότι το Κοινοβούλιο ε, δεν ε, συμφώνησε και δεν υποστήριξε την νομοθεσία ορισμένη. Όπως η Επιτροπή ε, Οικονομικών Υποθέσεων μιλούσε για 100% ατέλεια, όλοι δωρεάν άδειε. Αλλά δεν μπορεί κανείς αυτό να θεωρεί ότι το Κοινοβούλιο αποφάσισε ούτως. Το Κοινοβούλιο αποφάσισε άπαξ. Μπορεί να μην ήταν καλή η διαδικασία, αλλά ήταν η μόνη ε, ομάδα, η δική μας, που αμφισβήτησε τη διαδικασία. Όλοι οι άλλοι ήταν υπέρ. Το Κοινοβούλιο ψήφισε το Δεκέμβριο. Λοιπόν, και υπάρχει και η ημερομηνία και η διαδικασία για τη λίστα. Οπότε δεν μπορούμε να ε, κατηγορήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν το εφήρμοσε αυτό. Τώρα, το βασικό επιχείρημα κατά του ψηφίσματος είναι ότι δεν ελήφθη λέει υπόψη ε, η στάση των τρίτων κρατών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκαθάρισε τη θέση της όμως. Είπε ότι δεν υπάρχουν νομικά δεσμευτικές αποφάσεις άλλων βουλών. Και προεκλογικά μπορεί κανείς να εξαγγέλει διάφορα πράγματα ή στις προγραμματικές δηλώσεις. Αυτό όμως δεν είναι νόμος. Βλέπουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες πόσο κοστίζει μια προεκλογική εξαγγελία να την κάνει νομοθεσία. Το ξέρουμε αυτό και στην Ένωση. Καλά είναι οι προτάσει, καλέ είναι οι προθέσει, αλλά δεν είναι ακόμα νόμος. Και θα πρέπει να υπάρχει και μια ασφάλεια για τι επιχειρήσει, ε, για του εργαζομένου, για τι θέσει απασχόληση. Είναι σοβαρά αυτά τα πράγματα και δεν μπορούμε να βασιζόμαστε σε εξαγγελίε ή ε, προθέσει Και τελικά να αποκλίνουμε από τα όσα αποφασίζουμε. Επίσης είναι πολύ προβληματικό αυτό που λένε ορισμένοι συντάκτες του ψηφίσματος ότι η αποτελεσματικότητα δεν είναι παντού σε όλες τις τρίτες χώρες υπό όλες τις συνθήκες χειρότερη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί στη Βραζιλία ή στην Κίνα να έχουμε ένα εργοστάσιο χάλιβα που να είναι ε, όπως στην Ευρώπη, τα στάνταρ και οι προδιαγραφές. Εγώ όμως θα πρέπει να πάω στη χώρα μου στην ιδιαίτερη πατρίδα μου και να πω στους εργαζομένους ότι εάν είναι η ίδια αποτελεσματικότητα και δεν βλάπτει το κλίμα, μπορούν να μετακατασταθούν οι άνθρωποι, να πάνε εκεί αφού δεν ρηπαίνουν παραπάνω. Άντε να το εξηγήσει αυτό στον κόσμο, ότι δεν βλάπτει το περιβάλλον, αλλά βλάπτει τους εργαζομένους μας που θα απολυθούν. Και το κόστος των μεταφορών, όταν δεν παράγεται το χάλιβα στην Ευρώπη, αλλά εισάγεται. Και έχουμε και το κόστος των μεταφορών, λοιπόν, που είναι και πάλι επιβαρυτικό για το περιβάλλον. Λοιπόν, ε, ας μην το μεταχειριζόμαστε τόσο πολύ αυτό το επιχείρημα. Και μπορεί κάπου στον κόσμο να βρει ένα χαλιφουργείο Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είναι ε, ίδιων προδιαγραφών και τι θα γίνει, λοιπόν, θα βγάλουμε 100% φυρμάνι για ε, πληστηριασμό των αδειών. Ακούστηκε και το επιχείρημα ότι είμαστε πολύ φιλόδοξοι. Κοιτάξτε, ποια είναι τα ε, γεγονότα. Τώρα έχουμε ένα σύστημα εμπόριου που εκπομπών που λειτουργεί χωρίς πληστηριασμούς. Η Γερμανία, η η Αγγλία στα θερμοελεκτρικά εργοστάσια έχουν ήδη 10% στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος και το 2013 θα περάσουμε στο 100% στους πληστηριασμούς και στις χώρες κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης λίγο αργότερα. Δηλαδή θα υπάρχουν πολύ περισσότεροι πλέον πληστηριασμοί και δεν έχουμε υπερβολική ε, διάθεση δικαιωμάτων. Στην αρχή ήταν πάρα πολύ κακέ οι επιδόσει. Τώρα κάποιοι επικρίνουν το benchmark, τη συγκριτική αξιολόγηση. Αν δεν είχαμε θεσπίσει από την αρχή θα είχαμε προχωρήσει πολύ περισσότερο στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγή. Το benchmarking λοιπόν δεν είναι κατά του περιβάλλοντο, είναι θετικό στην περιβαλλοντική πολιτική ω μέσο. Και τελευταίο το επιχείρημα με τι Ηνωμένε Πολιτείε. Λοιπόν, εάν στι Ηνωμένε Πολιτείε άκουγε κάποιος τη σημερινή μας συζήτηση για τον κατάλογο αυτό του carbon leakage και το χρησιμοποιήσει ως επιχείρημα ότι εμείς υπαραχωρούμε στην περιβαλλοντική μας πολιτική, δεν μας βοηθάει. Γιατί αν θεωρούμε όλοι ότι δεν είναι φιλόδοξη η δική μας προσπάθεια, τι να πει και η γερουσία και τι να πει και η Βουλή των αντιπροσώπων. Ε, ας το αντιγράψει όπως είναι αφού έχουμε στόχο 20% να γίνει 30%, 100% πληστηριασμοί για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και ε, το benchmarking ε, στην μεταποιητική βιομηχανία να παίρνει την άδεια μόνο όποιος έχει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Αυτό σας φαίνεται ε, χαμηλή φιλοδοξία. Ε, τότε αγαπητοί γερουσιαστέ και αντιπρόσωποι των ΗΠΑ, αντιγράψτε το και να δείτε τι τεράστια επιτυχία θα είναι η Κοπενχάγη. Εμείς έχουμε στόχους, έχουμε την προθυμία να συνεχίσουμε και όποιος θέλει να μας ακολουθήσει, δεν χρειάζεται να μας κατηγορεί, ας μας ακολουθήσει. Έχουμε και αξιολόγηση και όχι μόνο 100% πληστηριασμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ η Κορίν Λεπάζο. Κύριε Πρόεδρε, δεν πιστεύω πως ε, κάποιος εδώ αμφισβητεί τον κατάλογο που έχουμε ψηφίσει. Αυτό δεν το άκουσα από κανένα. Πρώτη μου παρατήρηση αυτό. Δεύτερη παρατήρηση. Δεν πιστεύω ότι οποιοδήποτε έχει αμφισβητήσει τους στόχους που έχουμε και τους οποίους έχουμε ψηφίσει στο πλαίσιο αυτής της νομοθεσίας. Τι θέλουμε. Θέλουμε να δούμε αν ο πρώτος κατάλογος που μας παρουσιάστηκε και κανείς, όπως είπαμε, δεν τον αφισβήτησε ούτε και το γεγονός ότι η Κομισιόν έκανε τη δουλειά της, παρουσιάζοντάς μας αυτό το κατάλογο στις προθεσμίες που τις είχαμε θέσει. Δεν είναι θέμα λοιπόν αυτό. Το πραγματικό θέμα είναι αν θα μπορέσουμε ή όχι να πετύχουμε τους γενικούς στόχους που έχουμε θέσει. Και στο ψήφισμα, αυτό ακριβώς θέλουμε να γνωρίζουμε, αν έχοντας μία τόσο ευρεία αντίληψη των αποκλεισμένων τομέων, μήπως καθιστούμε σχεδόν αδύνατον την πιθανότητα να απαντήσει κανείς και να ανταποκριθεί στους ε, τόσο δεσμευτικούς στόχους που έχουμε θέσει. Ε, αυτό είναι το θέμα. Δεν νομίζω πως υπάρχει άλλο ζήτημα. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το θέσουμε, όχι γιατί είμαστε βέβαιοι ότι θέλουμε ότι αυτό μάλλον θα βλάψει την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Κανεί δεν το επιθυμεί αυτό, είναι αυτονόητο. Αλλά η προετοιμασία της Κοπενχάγης είναι πολύ καλό παράδειγμα για κάτι τέτοιο, αλλά γιατί το να θέτουμε στόχους διαρκώς είτε πιο ελαστικούς είτε πιο επιθετικούς για να τα, τους πετύχουμε ε, είναι ο καλύτερος τρόπος για να μην τα καταφέρουμε τελικά. Πιστεύω λοιπόν ότι πραγματικά ο κατάλογος αυτός είναι εξαιρετικά μακρύς και ότι θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση με την Κομισιόν και χαίρομαι και θα μπορέσουμε να θέσουμε το, το ερώτημα αυτό στον κύριο Δήμα σε λίγο ότι αυτό το θέμα που τελικά καλύπτει το, 70-90 το, των ευρωπαϊκών εταιριών, αν τελικά ξεπερνά αυτή την αρχή της βάσης, ε, τη βασική μάλλον αρχή. Ε, πιστεύω πως ε, θα πρέπει να είμαστε αντίθετοι, γιατί αν όντω θέλουμε να προχωρήσουμε προς ένα σύστημα το οποίο είναι σύστημα <laughs> ευραίων εξαιρέσεων, καταρχήν θα, θα θα, θα, θα στρεβλώσουμε τελείως την αγορά του άνθρακα που δεν το χρειάζεται κάτι τέτοιο και δεύτερον θα βρεθούμε σε αδυναμία να ανταποκριθούμε στους στόχους ακόμα και του 20% που θέσαμε για το 2020 και γι' αυτό το λόγο ακριβώς προσωπικά εκτός και αν ο κύριος Δήμα μας πει κάτι το εξαιρετικό θα υποστηρίξω αυτό το ψήφισμα. vielen Dank. Ε, ευχαριστώ πολύ. Κατρίν Σουγιέ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ ίσω να περιτεύω αυτά που θα πω σε σχέση με τα όσα υπόθηκαν μέχρι στιγμή, αλλά ήθελα να υποστηρίξω το σχέδιο πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό για του εξή τρει λόγου. Ο πρώτο είναι ότι η πρόταση τη Κομισιόν ε, σέβεται μια συνένεση και αυτό υπόθηκε επανειλημμένω ότι ο που εκτίθεται, ε, η λίστα των τομέων μάλλον που εκτίθεται στις διαρροέ Αφρικα είναι, ε, είναι κατάλογος ο οποίο έχει συνταχθεί με πυρογνώμονες των κρατών μελών, εμπειρογνώμονε τη βιομηχανία, Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι πίσω από τι επιχειρήσει υπάρχουν θέσει απασχόληση επίση Δεύτερον, αυτή η πρόταση εισάγει μία, μία έντονη προσπάθεια μείωση ε, των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Η συμπερίληψη ενό τομέα εδώ στον κατάλογο δεν σημαίνει πω θα εξαιρείται από την προσπάθεια μείωση των εκπομπών. Οι ευρωπαϊκέ εταιρείε ε, είναι υποχρεωμένε να μειώσουν τι εκπομπέ του, ακόμα και αν δεν υπάρχουν ανταγωνιστές ε, αντίστοιχοι στις ε, χώρες εκτός Ένωσης ε, και εντός Ένωσης. Είμαστε κάπως αισιόδοξοι σε σχέση με την Κοπεχάγη. Δεν χρειάζεται, δεν υπάρχουν λόγοι για να αποτύχει. Και όπως προβλέπει και η ίδια η οδηγία, το συζητήσαμε προηγουμένως το 10β παράγραφος 1, ότι δηλαδή ο κατάλογος μπορεί να μεταβληθεί από το φως των διαπραγματεύσεων των διεθνών και σε σχέση με το πώς θα περιοριστούν οι εκπομπέ των αερίων του θερμοκηπίου μετά από τη Διεθνή Συμφωνία. Εγώ θα είμαι κατά λοιπόν τη υιοθέτηση αυτού του ψηφίσματος. Ωραία, Κάρλ Σλίτερ. Να πω στους συναδέλφους μου ότι συμφωνούμε σε όλα αυτά, συμφωνήσαμε μάλλον και άρα στην ουσία λένε γιατί να ταράξουμε τα νερά τώρα, να τα ταράξουμε εγώ σα λέω ότι η Κομισιόν δεν κάνει αυτό που έπρεπε να κάνει. Αν θέλετε ένα επίσημο νομικό επιχείρημα αυτό πρέπει να κάνουμε. Αν, υπά, αν υποτίθεται ότι θέλουν να μειωθούν οι εκπομπέ και εκτό Ευρώπη. αν υποτίθεται ότι λαμβάνουν υπόψη τι δεσμεύσει των άλλων χωρών, τότε είναι πολύ σκόπιμο για το ποιε, το να ασχοληθούμε με το ποιες βιομηχανίες θα συμπεριληφθούν σε αυτόν τον κατάλογο. Γιατί Αν κάνουμε λάθος, αυτό θα υποσκάψει μια διεθνή συμφωνία. Γιατί εμείς θα βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις μας να ξεφύγουν από ένα μεγάλο κομμάτι της δικής τους ε, οικονομικής ευθύνης και άρα αν θα, θα, θα, υπάρξει, θα, αποτύχει διεθνώς η, η συμφωνία. και θα χάσουμε κάθε ωφέλεια από ένα τέτοιο πρόβλημα. Οι εταιρείε που δεν θα είναι στον κατάλογο θα είναι αυτές που θα πληρώσουν περισσότερο για τις ε, πληρωτές άδειες και τις οποίες δεν χρησιμοποιούν. βασίζεται στο 10% του πιο αποτελεσματικού μέσα στο 2007 και 2008. Θα έχουμε δηλαδή ένα ποσοστό φυσικής αποδοτικότητας ε, ε, που σημαίνει πως πάνω από το 10% θα πάρει δωρεάν άδεια για το 2013-2014 θα έχουν την ποσόστοση. Θα καταλήξουμε σε μια κατάσταση όπου πολλές εταιρείε δεν θα προβούν στις απαραίτητες επενδύσεις, δεν θα δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης. Συγγνώμη κύριε Ρώση, αλλά το επιχείρημά σας είναι σαθρό. Εάν δεν γίνονται επενδύσεις δεν δημιουργούνται και θέσεις απασχόλησης και άρα εγώ είμαι πολύ απογοητευμένος με τη συμφωνία που κάναμε. Δεν είμαι ευχαριστημένο με το νομικό κείμενο επί το οποίο βασίζεται. Εγώ θα προτιμούσα ένα πολύ πιο, πιο ισχυρή οδηγία. Ο καθένα δηλαδή πρέπει να πληρώνει για τις ε, ποσοστώσεις τους εγώ έχασα σε μεγάλο βαθμό. Αλλά ένα μικρό πραγματάκι που κερδίσαμε ήταν ότι δεν μπορούμε να το δίνουμε δωρεάν σε όσους γίνεται περισσότερο χωρίς να σκεφτόμαστε τις επιπτώσεις για τις άλλες χώρες. Και εκεί νομίζω πως εν γέννη όσοι είναι ευχαριστημένοι με το συμβιβασμό που φτάσαμε θα έπρεπε να σκεφτούν και να δεχτούν και εκείνο το φίλο εκεί που έχει μείνει για του περιβαλλοντολόγου και τουλάχιστον συγκρίνουμε και τους, ε, αυτού μα με άλλου και να μην παραβλέψουν αυτή τη νίκη που είχαμε. Γιατί πολλοί κόσμοι που είναι φιλικός με το περιβάλλον θέλει, θέλησε να τα βελτιώσει τα πράγματα και το πέρασε αυτό και τώρα ορισμένοι θέλουν απλώ να γνωρίσουν τη συμφωνία. Απαράδεκτο. Γι' αυτό και σα ζητώ να υπερψηφίσετε αυτό το ψήφισμα αν όχι, δεν ε, υποστηρίζετε την συμφωνία την οποία εσείς ήδη υπερψηφίσατε. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε νομικίστικα επιχειρήματα, ε, θα πρέπει να υπερψηφίσετε αυτό το κατάλογο για να διορθωθεί αυτό σύμφωνα με την ε, ε διαπραγμάτευση που κάναμε ανάμεσα στα όλα τα θεσμικά όργανα. Τώρα για, το, για τον κύριο Κάλαναν δεν είδα διαβάζοντας την έκθεση της UNESCO το κατά πόσο οι ευρωπαϊκές το πώς είναι μάλλον οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να είναι πιο αποτελεσματικές όσον αφορά την παραγωγή λιπασμάτων, ούτε καν στην παραγωγή μουσικών οργάνων, ούτε καν στην παραγωγή βουρτσών. Αν συγκριθούμε με τους άλλους λοιπόν, πολλοί τομείς μας θα εξαφανιστούν, πράγμα το οποίο θα είναι σωστό και σύμφωνο με τη συμφωνία. Αν επιμείνουμε στη συμφωνία του Δεκεμβρίου, ε, θα πρέπει να υπερψηφίσουμε αυτό το ψήφισμα. Yeah. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να εκβιάσουμε κανέναν εδώ στην Επιτροπή μα. Ε, να πούμε δηλαδή ότι όποιο δέχεται τον κατάλογο προστατεύει το περιβάλλον, ενώ οι υπόλοιποι όχι. και να πούμε ότι οι υπόλοιποι σύμφωνα με το άρθρο 10α είναι κακοί προστάτες του περιβάλλοντος. Ε, θα καλούσα τον ε, Καλ Σλίτερ να διαβάσει σωστά το άρθρο 10α και να δει αν τα κριτήρια που αναφέρονται εκεί πληρούνται ή όχι. Θα ακούσουμε όμως και την Κομισιόν. Νομίζω σιγά σιγά ότι θα πρέπει να κλείσουμε τη συζήτηση, διότι βλέπω δευτερολογίες. Πέντε έχω ακόμα στον κατάλογο των ομιλητών. Ε, θα παρακαλούσα την κυρία Σλίγενπερτ να μας πει τι συνέβη, διότι συμμετείχε στην ε, σύνταξη του καταλόγου. Euh, Κύριε Σπερνιό, ε, πρέπει να σας πω ότι αισθάνομαι πάρα πολύ άβολα από την αρχή της συζήτηση. αυτής. Έχω την εντύπωση ότι θα έρθει τώρα ο Επίτροπος στις 11 η ώρα ο κύριος Δήμας να τον ακούσουμε. Και αλλά ακούω ε, να παίρνουν πολιτική θέση εδώ διάφοροι χωρίς να επανερχόμαστε στην νομοθετική δουλειά που κάναμε στην προηγούμενη θητεία. Και εγώ, όπως και άλλοι, είμαι νέος ευρωβουλευτής εδώ Αλλά μελετώντας το φάκελο, έχω ανάγκη να το διαβάσω και να αναρωτηθώ. Τι έγινε, στην προηγούμενη θητεία λήφθησαν κάποιες αποφάσεις τώρα, αυτό είναι πρόοδος, είναι επίτευγμα, μπορούμε να προχωρήσουμε σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση με το παρελθόν, είναι βελτίωση. Άκουσα τη Λίντα Μακάβαν ε, που συμμετείχε στον τριμερή διάλογο εκπροσωπώντας μας και θα ακούσω και τον Επίτροπο. Euh, Για να αποκομίσω άποψη κι εγώ και να δω πώς θα ψηφίσω τελικά. Πάντως έχει σημασία ε, η απόφαση αυτή να ληφθεί μετά από ε, σωστή αξιολόγηση ανάλογα με το στόχο μας. Τι επιδιώκουμε, σε τι αποσκοπούμε και υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο, όπως το έχουμε θεσπίσει και όπως ε, θέλουμε να είναι, για να προστατευτούμε από την υπερθέρμανση του πλανήτη. Και επίσης κάτι άλλο που πρέπει να ρωτήσουμε τον Επίτροπο είναι τι θα γίνει με αυτόν τον κατάλογο. Και εμένα μου φαίνεται μακροσκελέστατος ε, σε σχέση με το ιδεώδη που θα επιθυμούσα για την καταπολέμηση. Αλλά αυτός ο κατάλογος είναι απόλυτος. Ε, είναι οριστικός. Μετά την Κοπεχάγη δεν μπορούμε να τον αναδιαμορφώσουμε ανάλογα με τη βούλησή μας. Αν έρθει αύριο κάποιος και μου πει ότι μπορεί να αλλάξουν αυτά τα πράγματα, δεδομένη τη ισχυρή ε, βούληση που έχουμε για το περιβάλλον, δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην εξακολουθήσουμε να εργαζόμαστε σε αυτή τη νομοθετική διαδικασία. Και τέλος, καμιά φορά ακούω αντιφατικά πράγματα από τους συναδέλφους που αρνούνται ε, τους δασμούς στα σύνορα της Ευρώπης και ταυτόχρονα μας λέγουν ότι ο κατάλογος αυτός είναι πάρα πολύ μακρύς και θα πρέπει κάπου να έχουμε ε, άλλη πολιτική πιο ισχυρή υπέρ του περιβάλλοντος. Ε, όπως και να το κάνουμε είναι κάπως αντιφατικά αυτά. Δηλαδή, ε, καλό είναι να είμαστε ρεαλιστές, αλλά να έχουμε και τη βούληση στα πλαίσια της ε, νομοθετικής μας ε, προσπάθειας που αποφασίσαμε πέρσι και μάλιστα συν αποφασίσαμε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ριβελίνη. Grazie Presidente. <clears throat> È un voto importante, difficile e sono oggettivamente είναι πολύ σημαντική και δύσκολη ψηφοφορία και πραγματικά είμαι αναποφάσιστο. Ο συνάδελφο Ρώση έχει δίκιο. Η Ευρώπη, για να κάνουμε μια, σύγκριση, έχει μια πολιτική ε, περιβαλλοντική που είναι ισχυρή με τους ε, αδύναμους και αδύναμη με τους ισχυρούς. Στα σύνορά μας ε, οι εκπομπές των επιχειρήσεων είναι εκτός κάθε λογικής και εδώ ε, μπαίνουμε σε μια, ένα πρόγραμμα και μια πολιτική, μια προοπτική που δεν θα έπρεπε να είναι ευρωπαϊκή μόνο, αλλά διεθνής. Και ε, μάλιστα δεν έχουμε χρησιμοποιήσει τι ευκαιρίες για να επιμείνουμε με στένος. Ε, την ίδια θέση και την ίδια στένος δεν έπρεπε να το δείξουμε όταν, για παράδειγμα, ορισμένα μεγάλα έθνη μπήκαν στον WTO χωρίς να κάνουν καμία υποχώρηση κανενό είδου ακόμα και στις περιβαλλοντικές πολιτικές. Και επίσης, ε, να σας πω και κάτι λίγο κακό. Είμαστε, υπάρχουν ε, επιχειρήματα μεγάλα λόμπι, τα με τεράστια λόμπι, πιο μεγάλα από την Ευρώπη. Πραγματικά είμαστε πεπισμένοι ότι ανησυχούν ε, για την ψήφο μας. Ή μήπως για αυτούς είναι, για τα μεγάλα λόμπι, ένα μέσο για να μπορέσουν να μεταφέρουν τις δραστηριότητε του στι χώρε του τρίτου κόσμου όπου το κόστο της εργασίας είναι πολύ πιο χαμηλό και βολικό και οι περιβαλλοντικές πολιτικές πολύ πιο χαλαρές. Βεβαίω, αυτό ισχύει για τα, για τα μεγάλα λόμπι ενώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυτή η ψηφοφορία μπορεί να είναι καθοριστική και εξαιρετικά αρνητική και η μεγάλη πλειοψηφία των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην Ιταλία είναι σχεδόν 90% οι επιχειρήσεις που είναι μικρές και μεσές για να ε, διαμαρτυρηθούν για την ευρωπαϊκή πολιτική που είναι ισχυρή με τους αδύναμους και αδύναμη με τους ισχυρούς και για να προστατεύσουμε αυτήν, ε, την, αυτές τις μικρές επιχειρήσεις που βρίσκονται στο έλεος της δικής μας ψηφοφορίας, της ψήφου μας χωρίς ε, κατάλληλη προστασία, εγώ θα καταψηφίσω. Ευχαριστώ κύριε Ριβελίνη. Τώρα έχουμε τον κύριο καμπράντι. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ε, λέει κύριο Γκαρμπράντη, είμαι και εγώ νέο μέλο στην Επιτροπή και με κάποια έκπληξη ακούω τη συζήτηση όλη. Έχω την αίσθηση ότι πολλά μέλη που έζησαν τη συζήτηση του 2008 έχουν ταμπουρωθεί σε κάποια χαρακόμματα και κάνουν συζητήσεις άστοχες και άκερες. Δεν συζητάμε τον κατάλογο αυτόν καθευτό, ούτε το νόημα του καταλόγου με τις εξαιρέσεις του. Αυτά τα έχουμε ε, ε, λήξει. Ε, είναι περσινά ξινά στα φιλιά. Δεν θα πρέπει να ξανανοίξει αυτή η συζήτηση. Αυτό που με εκπλήσει επίσης είναι το χρονοδιάγραμμα της λίστας. Ξέρω ότι ζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να φέρει τώρα την πρόταση, αλλά θα μπορούσαμε να ε, αναρωτηθούμε αν είναι τόσο ευτυχής η συγκυρία. Είναι σωστό να κυκλοφορεί ο κατάλογος αυτός τώρα τέτοιες ώρες. Μας ικανοποιεί, μας χαροποιεί. Εγώ ως φιλελεύθερος ε, ε, θέλω και θεωρώ πολύ σημαντικό να έχει ασφάλεια η βιομηχανία. Να ξέρει πού πηγαίνει, να ξέρει τι την περιμένει, να ξέρει τι μακροχρόνιες επενδύσεις μπορεί να κάνει. Ε, ποια ασφάλεια δίνουμε εμείς στην βιομηχανία καταρτίζοντας από τώρα ένα κατάλογο ε, ο οποίος μετά από ένα μήνα μπορεί να ανατραπεί μετά την Κοπεχάγη ή να αναθεωρηθεί. Τι θα σου πει η βιομηχανία. Ποιος θα πιστεί αν μπορείτε να με πείστε με επιχειρήματα ποια βιομηχανία θα βασιστεί σε αυτόν τον κατάλογο που μπορεί μετά από δύο μήνες να μην ισχύει καθόλου, να ανατραπεί εξ ολοκλήρου. Ε, δεν ξέρω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ίδια είναι ικανοποιημένη με αυτό το χρονοδιάγραμμα. Για λόγους λοιπόν χρονικούς εγώ ε, υποστήριξα το ψήφισμα και θα ξεκολουθώ να το υποστηρίζω και ε, θέλω να αποσυρθεί τώρα ο κατάλογος και μετά την Κοπεχάγη σε ανανεωμένη και αναθεωρημένη μορφή να επανυποβληθεί. Ευχαριστώ πολύ. Das Timing steht nur leider im Gesetz. Das äh, war nicht äh, zu, unserer, äh, zu unserem Wunsch. Aber... Δυστυχώς το χρονοδιάγραμμα το λέει ο νόμος. Δεν το είχαμε επιθυμήσει εμείς έτσι, αλλά το δεχτήκαμε. Γιολάντα Χίπνερ. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowni państwo, ja się przysłuchuję i... Κυρίες και κύριοι, Άκουσα τη συζήτηση, αλλά κατά καιρού μου φαίνεται ότι έχω παρεστήσεις. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αποτελούν πρόβλημα για μας. Μερικές φορές νομίζω ότι δεν καταλαβαίνουμε ότι αυτές οι επιχειρήσεις παρέχουν θέσεις απασχόλησης και οικονομική ανάπτυξη. Μιλάμε για, ευρωπαϊκές, για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις Σαν να τους δίνουμε κάτι δωρεάν. Οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να πληρώσουν τελικά το λογαριασμό, όχι οι Κινέζοι. Εάν θέλουμε οικονομική ανάπτυξη σε αυτή την εποχή οικονομικής κρίσης, θα πρέπει να σκεφτούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις μας. Δεν έχει νόημα να καθυστερήσουμε περαιτέρω τη διαδικασία. Θα πρέπει να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να επενδύσουν. να τις βοηθήσουμε κατά τη διάρκεια μιας διετίας ε, κατά την οποία θα προετοιμάζονται για την ανάπτυξη. Το νόημα δεν είναι η συζήτηση για το ποιο τομέα θα πρέπει να συμπεριληφθεί ή να αφαιρεθεί από τον κατάλογο. Έχουμε πολλούς τομείς που δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στη ζήτηση για τις νέες τεχνολογίες, διό... στην απέτηση για τις νέες τεχνολογίες, διότι δεν υπάρχουν αυτές οι νέες τεχνολογίες και δεν μπορούμε να επιβάλλουμε άπειρες υποχρεώσεις σε αυτές τις επιχειρήσεις. Θα μπορούσαμε να κάνουμε πάλι την η διασυζήτηση του χρόνου. Αλλά όπω το χωρούμε κύριε και κύριοι, θα πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε τη συζήτηση για το αν ο κατάλογο είναι καλό ή κακό, αν θα πρέπει να γίνει επαναξιολόγηση. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να φοβηθούμε το να λάβουμε μια απόφαση. Πριν να δώσω το λόγο στην κυρία Σλίνγκμπερ και η κυρία Σάτου Χάση ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Μία παρατήρηση προς τον κύριο Ζίμπερκ και άλλους που είπαν ότι ο κατάλογος αυτός σημαίνει ότι μόνο το 10% των επιχειρήσεων θα ε, λάβουν ε, ε, αυτομάτως άδειε. Το 10%, για το 10% ισχύει αυτό για τις πιο αποτελεσματικές ενεργειακά επιχειρήσεις. Αλλά σύμφωνα με την Επιτροπή το 77% θα συμπεριληφθεί στην ομάδα που θα υπόκειται στα ίδια κριτήρια. Πρόκειται δηλαδή για ε, τον μεγάλο όγκο των εκπομπών. Η δεύτερη και τελευταία παρατήρησή μου είναι η εξή. Πολλοί από εμά συμμετείχαμε σε διαπραγματεύσεις σχετικά με το shall ή το may. Το μπορεί ή πρέπει, αν η ρήτρα θα πρέπει να είναι δυνητική ή υποχρεωτική. Ξέρετε ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό σε ένα νομικό κείμενο. Στο συγκεκριμένο νομικό κείμενο λέμε shall. Πρέπει. Ο νόμος λέει ότι λαμβάνονται υπόψη οι δράσεις τρίτων χωρών. Δεν είναι θέμα λοιπόν πολιτικής αξιολόγησης της Κομισιόν, το αν θα το κάνει αυτό ή όχι. Αυτό όμως δεν γίνεται. όταν ε, λέμε ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η κατάσταση στις τρίτες χώρες. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να λαμβάνουμε μόνο υπόψη μας την ε, ενεργειακή αποτελεσματικότητα των χωρών αυτών, αλλά και τις υπόλοιπες συνθήκες και τίποτα από αυτά δεν λαμβάνεται υπόψη στους υπολογισμούς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Σλίνμπεργκ, πολλές ερωτήσεις ακούσατε. Υπόθηκε ότι δεν πληρούνται τα κριτήρια του άρθρου 10α. Η σύγκριση δηλαδή με παρόμοιες εγκαταστάσεις σε τρίτες χώρες. Δεν γίνεται ουσιαστικά. Δεύτερον, γιατί είναι τόσο μακρύς ο κατάλογος. Πρόκειται για αποτέλεσμα πολιτικής απόφασης. Ερωτήθηκε συγκεκριμένα γιατί συμπεριλαμβάνεται και ο τομέα του ίνου. Έχουμε και την ερώτηση την οποία θα πρέπει να απαντήσει και ο Επίτροπος κ. Δήμας. Πότε θα υπάρξει νέος κατάλογος μετά την Κοπεχάγη. Πώς θα συμμετάσχει το Κοινοβούλιο στην εκπόνηση του νέου καταλόγου. Και αν υπάρξει νέος κατάλογος, οι σχετικέ τροποποίησει θα γίνουν και προς τις δύο κατευθύνσεις, δηλαδή θα προσθεθούν ε, τομεί και θα αφαιρεθούν τομεί, διότι υπάρχουν ε, φόβοι απλά να προσθεθούν τομεί. Με ποια βάση λοιπόν θα γίνουν ε, οι κατάλογοι αυτοί και τι στόχους έχετε μετά την Κοπεχάγη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μερικές διευκρινήσεις από τη δική μας πλευρά. Ε, φυσικά θα αναφερθεί στο θέμα και ο Επίτροπος. Καταρχήν, σημαντικό είναι από την πλευρά μας να τονίσουμε ότι το σχέδιο απόφασης ε, στόχο έχει το ε, μονομερές ε, πρόγραμμα μειώσεων 20%. Θα γίνει επαναξιολόγηση μετά την Κοπεχάγη. Αυτό αναφέρεται στο 10β παράγραφος 1. Και η Κομισιόν θα πρέπει να υποβάλει την αξιολόγησή της ε, μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2010, ε, συνοδευόμενη από ε, σχετικές προτάσεις. Θα αναθεωρηθεί ο κατάλογος υπό το φως των διαπραγματεύσεων για την προστασία του κλίματος, των διεθνών διαπραγματεύσεων. Και Οποιαδήποτε αποτελέσματα θα περάσουν από τη διαδικασία της ε, συναπόφασης, θα, θα συναποφασιστούν δηλαδή από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Θα ήθελα να τονίσω ότι η πρόταση απόφασης ε, νομικά στέκει. Γιατί? Διότι η Κομισιόν έχει ακολουθήσει πιστά τις διατάξεις της οδηγίας στη διαδικασία αυτή και τα κριτήριά τη όπω αυτά υιοθετήθηκαν πέρσι. Επίσης, σέβεται η Κομισιόν την προθεσμία που συμφωνήθηκε πέρσι. Αυτό δεν συμπεριλαμβανόταν στην πρόταση τη Επιτροπή. Η Επιτροπή διαφωνούσε με την προσέγγιση αυτή. Εμεί πάντα θεωρούσαμε ότι ο κατάλογο αυτό θα πρέπει να υιοθετηθεί μετά την Κοπεχάγη, αλλά συμφωνήθηκε αυτό μεταξύ ε, Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Σεβόμαστε λοιπόν την απόφαση αυτή. Όσον αφορά τα διάφορα κριτήρια και την ανάλυση του τι κάνουν οι τρίτε χώρε. Ε, το 10α παράγραφος 18 λέει ότι ο κατάλογος ε, που αναφέρεται στο άρθρο 13 θα συντάσσεται λαμβάνοντας υπόψη και εδώ έρχεται ένα σημαντικό σημείο, όπου είναι διαθέσιμα τα σχετικά δεδομένα. Και δύο πράγματα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Ο βαθμός στον οποίο οι τρίτες χώρες που αντιπροσωπεύουν ε, αποφασιστικό κομμάτι της ε, διεθνούς παραγωγής ε, σε κάποιους τομείς που θεωρείται ότι μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαρροής άνθρακα. Το αν αυτές οι χώρες δεσμεύονται να μειώσουν τις εκπομπές αερίων και δεύτερον θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη την ενεργειακή αποτελεσματικότητα των εγκαταστάσεων που βρίσκονται στις χώρες αυτές. Στι χώρες αυτές δηλαδή που δεσμεύονται να μειώσουν τις ε, εκπομπέ ε, των ε, αερίων του θερμοκηπίου και που και που αποτελούν σημαντικό, που αντιπροσωπεύουν σημαντικό μέρο τη ε, διεθνού παραγωγή. Η Επιτροπή λοιπόν έχει λάβει υπόψη τη στα κριτήρια αυτή. Μόνο η Νορβηγία, η Ισλανδία και η Ελβετία έχουν δεσμευτεί να μειώσουν ε, τα αέρια των θερμοκηπίων, τι εκπομπέ αερίων του θερμοκηπίου στου ε, σχετικού τομεί. Οι χώρε αυτέ, ακόμα και μαζί, δεν αντιπροσωπεύουν αποτελεσματικό κομμάτι τη διεθνού παραγωγή στου εν λόγω τομεί. Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα την ενεργειακή αποτελεσματικότητα. Η Κομισιόν λέει ότι δεν υπάρχουν τα απαραίτητα στοιχεία λόγω της μη συγκρισιμότητας των στοιχείων και της έλλειψης διεθνών στοιχείων. Ε, και καθότι η το σχέδιο απόφαση λέει ότι μόνο η Νορβηγία, η Ισλανδία και η Ελβετία έχουν δεσμευτεί να μειώσουν τι εκπομπέ αερίων του θερμοκηπίου και δεν, ε, δεν αντιπροσωπεύουν αποφασιστικό κομμάτι τη διεθνού παραγωγή, ε, δεν έχει νόημα να αξιολογήσουμε την, ε, την ενεργειακή αποτελεσματικότητά του. Στι περιπτώσει λοιπόν που εξετάσαμε τα στοιχεία αυτά, ήταν αυτά που, απαιτείται σύμφωνα με την οδηγία. Κάναμε μία μελέτη σχετικά με την ε, ενεργειακή αποτελεσματικότητα διεθνώς ε, με βάση τα ε, στοιχεία που υπάρχουν. Ωστόσο, τα στοιχεία αυτά δεν είναι αρκετά αξιόπιστα ώστε να, να μπορούν να ληφθούν υπόψη και να αλλάξουν τον τρόπο σύνταξης του καταλόγου. Η σχετική μελέτη θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα μας. στο σχέδιο ψηφίσματος της Επιτροπής ε, Περιβάλλοντος ε, για τα συμπεράσματα της Κοπεχάγης αναφέρεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μόνος περιφερειακός φορέας ε, του κόσμου που έχει αναλάβει υποχρεώσεις ε, σχετικά με την ε, μείωση αερίων του θερμοκηπίου έχοντας υιοθετήσει το κλιματικό πακέτο. Η Κομισιόν συμφωνεί με αυτό και περιμένει από τις τρίτες χώρες να δεσμευτούν να μειώσουν τα αέρια του θερμοκηπίου στην Κοπεχάγη. Η απόφαση ε, αντικατοπτρίζει την κατάσταση πριν ε, αναλυθούν τέτοιες υποχρεώσεις και γι' αυτό λέμε ότι η απόφαση θα αναθεωρηθεί υπό το φως των αποτελεσμάτων της Κοπεχάγης. Η Κομισιόν δηλαδή ακολούθησε κατά γράμμα τις διατάξεις αυτές και υπέβαλε την πρότασή της ώστε να μπορεί ε, τυπικά να εγκριθεί πριν το τέλος της χρονιάς. Έχουν γίνει πολλές παρατηρήσεις σχετικά με την δημοπράτηση ως προτινόμενη μέθοδο. Θα ήθελα να τονίσω ότι η δημοπράτηση συνεχίζει να αποτελεί τον κανόνα στην αναθεωρημένη οδηγία για το σύστημα εμπορίας εκπομπών. Ωστόσο, έχουν συμφωνηθεί κάποιες ε, διατάξεις για την ε, μείωση των αερίων και μπορεί να δοθούν ελεύθερες άδειες σε κάποιες επιχειρήσεις μέχρι το τέλος της επόμενης χρονιάς. Θα επανέλθουμε στην Επιτροπή σας με τα σχέδια προτάσεών μας για τα σχετικά benchmark, για τα σχετικά σημεία αναφοράς. Δεν υπάρχει όμως καμία πρόθεση να εξαιρεθούν οι τομείς που βρίσκονται στον κατάλογο των, της Κομισιόν. Μιλάμε μόνο για τις επιχειρήσεις ε, με απόδοση που ανταποκρίνεται στο στα benchmarks, δηλαδή ε, μιλάμε για το 10% των επιχειρήσεων. Ε, αυτές μπορούν να λάβουν δωρεάν ε, άδειες. Επειδή όμως δεν γνωρίζουμε ακόμα τα benchmarks, δεν μπορούμε να ξέρουμε το ακριβές ποσοστό του, της βιομηχανίας που θα καλύπτεται από το σύστημα αυτό. Το 77% δεν είναι σωστό. Αυτό αναφέρεται στο σύνολο του καταλόγου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι επιχειρήσεις στον κατάλογο θα λάβουν το 100% των ε, ε, εκπομπών τους ε, δωρεάν. Αυτό θα γίνει μόνο μέχρι το, μέχρι το επίπεδο του benchmark. Όσον αφορά τον τομέα του ίνου, ακολουθούντας τις διατάξεις και τα πολύ σαφή κριτήρια της οδηγίας, Θα πρέπει να φροντίσουμε οι ε, καταστάσεις εσωτερικής καύσης να καλύπτονται από την ε, οδηγία. Δηλαδή, οι εγκαταστάσεις που ακολουθούν τη διαδικασία αυτή καλύπτονται από την οδηγία για το σύστημα εμπορίας εκπομπών. Αυτό ισχύει για τον τομέα του ίνου και πολλούς άλλους τομείς που περιλαμβάνονται στο κατάλογο. Δηλαδή, οι τομείς αυτοί συμπεριλαμβάνονται λόγω, της, ε, λόγω των εγκαταστάσεων εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιούν θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας τα κριτήρια. Όταν εξετάζουμε δηλαδή το κατάλογο του ΙΝΟΥ, τα στοιχεία δείχνουν ότι ε, ε, έχουν άνοιγμα ε, εμπορικό προς τις τρίτες χώρες πάνω από 30%. Η Επιτροπή έκανε τη σχετική ανάλυση και με βάση τα κριτήρια αυτά συμπεριλήφθηκε ο, ο τομέας του ίνου στον κατάλογο. Όσον αφορά την εσωτερική καύση, ε, για την ε, παραγωγή ενέργειας δεν θα, υπάρξει, ε, δεν θα υπάρξουν δωρεάν άδειε για κανέναν. Μπορεί όμως να υπάρξει κάτι τέτοιο για την παραγωγή θερμότητας. Σε, κάποιο, σε περίπτωση λοιπόν που ένας το, που υπάρχει μια εγκατάσταση εσωτερικής καύσης για την η παραγωγή ε, θερμότητας μπορεί να ε, συμπεριληφθεί στο σύστημα. Είναι πολύπλοκο το σύστημα, δεν μιλάμε όμως για 77% όλων των ε, εκπομπών. Αυτό θα το δούμε με βάση τα benchmarks και σίγουρα δεν υπάρχει εξαίρεση όλων των τομέων αυτών από το σύστημα της δημοπράσης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Yeah. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σουμπέρκ για τις απαντήσεις σας αυτές. Όπως είπαμε, θα ψηφίσουμε για το θέμα αυτό μετά τη συζήτηση με τον Επίτροπο κύριο Δήμα, που θα έρθει να δώσει και εκείνο εξήγηση. Προτείνω λοιπόν να περάσουμε στο επόμενο θέμα της μέρης της διάταξης, που είναι το υπαριθμόν 8. Ορίστε, διαδικαστικό η Λίντα Μακέβαν. Θέλω να πω μόνο ότι η δική μου ομάδα θέλει να ζητήσει το εξή. Να ακούσουμε τον κύριο Δήμα και μετά διάλειμμα 5 λεπτά για να εκτιμήσουμε, ε, να σκεφτούμε τι θα μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν μπορείτε να το δεχτείτε, πέντε λεπτά διάλειμμα για να συντονιστούμε και μετά ψηφίσουμε. Το κατανοώ, αλλά μου φαίνεται δύσκολο να διακόψουμε 12 και 4. Πού θα μαζέψει τον κόσμο και ξανά στις 12.30 να ψηφίσει. Δεν ξέρω, είναι κυρίαρχη όμως η Επιτροπή. Έχετε παρατηρήσει αυτό? Ο Κρυς Θα συμφωνούσα με τη Λίντα Μακάβαν, πρόεδρε. Έχουμε κάνει συζητήσεις και στις ομάδες μας. Εχθές το βράδυ διχαστήκαμε. Είπαμε ειδικά να ακούσουμε τον Επίτροπο και πέρα από τα όσα ακούσαμε, ε, αυτό που θα μας πει θα είναι αποφασιστικά για να διαμορφώσουμε τη στάση μας στην ψηφοφορία. Πέντε λεπτά διάλειμμα, να είμαστε βέβαιοι ότι θα είναι ενωμένε οι ομάδες. Πρόεδρε, λέει η κυρία Μακέβαν, δεν είπα να εξαφανιστούμε. Πέντε λεπτά να μείνουμε στην αίθουσα. Το έχουμε ξανακάνει πολλέ φορέ να συνεννοούνται οι ομάδε πριν την ψηφοφορία. Δεν είναι πρόβλημα. Ο κύριο Σόνικ. Νομίζω ότι ακούσαμε όλα τα επιχειρήματα. Εγώ δεν πιστεύω ότι ο κύριος Δήμας θα ακομίσει τίποτα καινούριο και δεν νομίζω χρειάζεται καμία διακοπή πριν την ψηφοφορία. Εντάξει, έτσι λοιπόν θα διακόψουμε. 5-10 λεπτά μετά τις 12 και 4, έτσι και μία ψηφοφορία είναι υπέρ ή κατά. Μέχρι τις 12.30 θα έχουμε προλάβει να την κάνουμε. Αλλά παρακαλώ μην εξαφανιστείτε να μην μας διαλυθεί η Επιτροπή στις 12 και 4. Λοιπόν, γύρω στις 12 και 4, εν πάση περιπτώσει, 5-10 λεπτά διάλειμμα να κανονίσουμε την πορεία μας οι ομάδες. Ωραία. Πάμε τώρα στο 8. Είναι έκθεση κυρίας Ρόσπαχ για τη Σύμβαση Προστασίας του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος στο Βόρειο Ανατολικό Ατλαντικό, άλλος πως ΟΣΠΑΡ παραρτήματα που αφορούν την αποθήκευση ρευμάτων οδιοξιδίου του άνθρακα σε γεωλογικού σχηματισμούς. Η συγγήτρια έχει να μας πει τίποτα για τις τροπολογίες και ποιες συνιστά. Η κυρία Ρόσμπαχ, παρακαλώ. Ο Έλληνας συνάδελφος Κρήτων Αρσένης έχει υποβάλει μια πολύ καλή τροπολογία που ξεκαθαρίζει την κατάσταση. Δεν ξέρω. Ε, θα ήθελα να στηρίξω απόλυτα την τροπολογία αυτή Κάποιοι επιστήμονες με τους οποίους μίλησα μου είπαν ότι είναι ε, πολύ καλή λύση αυτή εφόσον δεσμευτεί ε, το διοξίδιο του άνθρακα ε, υπογείως. Ωστόσο μου είπαν ότι απαιτούνται πέντε ενότητες ενέργειας για να αποθηκευτεί μία ενότητα διοξίδιο του άνθρακα. Θα πρέπει δηλαδή να συμπιεστεί σε υγρή μορφή το διοξίδιο του άνθρακα για να αποθηκευτεί στο υπέδαφος ε, και το ερώτημα είναι μήπως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα που θα απαιτούσε κάτι τέτοιο για καλύτερες λύσεις. Ε, αυτή τη στιγμή βέβαια θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτό που έχουμε μπροστά μας. Θα ήθελα λοιπόν να συμφωνήσω με τις τροπολογίες του Κρήτονα. Μακροπρόθεσμα όμως θα πρέπει να βρούμε καλύτερες λύσεις από αυτήν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ο Κρις Ντέβις που είναι εισηγητής για την οδηγία αποθήκευσης, δέσμευση και αποθήκευση του διοξιδίου του άνθρακα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Τώρα έχω την ευκαιρία να κάνω διαφήμιση για το σεμινάριο που κάνω το μεσημέρι τώρα ε, για τη δέσμευση και αποθήκευση. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα ελάτε στις 12.30 θα έχουμε εκπροσώπους Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Μεταφορών και Ενέργειας. Θυμάμαι την επιφυλακτικότητα που είχαμε όταν πρωτοδιαβάσαμε αυτή την ιδέα. Δηλαδή, να παίρνουμε διοξίδιο του άνθρακα ε, από τα εργοστάσια και να το θάβουμε πολύ βαθιά ε, μέσα στους βράχους. Μίλησα όμως με ε, ειδικού στην Κίνα που μας είπανε ότι αυξάνεται πολύ η χρήση ορυκτών καυσίμων. Ακόμα και αν αυξηθούν δραματικά οι ανανεώσιμε πηγές ενέργειας τα επόμενα 20-30 χρόνια, δεν πρόκειται να φτάσει γιατί αυξάνεται η ζήτηση. Οπότε τα ορυκτά καύσιμα θα χρησιμοποιηθούν πολύ εντατικά τι επόμενε δεκαετίε και θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να περιορίσουμε τι εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα από τα ορυκτά καύσιμα. Όταν συζητήσαμε αυτή την οδηγία για την αποθήκευση γεωλογικού σχηματισμού, πριν από 1,5 χρόνο περίπου εδώ, αν θυμάμαι για πρώτη φορά και οι περισσότεροι βουλευτές που μίλησαν ήταν είτε εχθρικοί σε αυτή την ιδέα, είχαν πάρα πολύ σοβαρέ επιφυλάξεις. Έξι μήνες μετά όμως υπερψηφίσαμε την οδηγία και ε, όταν ήρθε το ETS βάλαμε και μία πρόβλεψη ε, για χρηματοδότηση για προγράμματα επίδειξης από τα χρήματα που περισσεύουν από το ETS. Το Κοινοβούλιο ανέλαβε την πρωτοβουλία και έπεισε και τους υπουργούς στο Συμβούλιο πέρσι. Έχουμε λοιπόν ένα καλό ιστορικό. Ε, στην αρχή είχαμε μια επιφύλαξη, αλλά τελικά να γνωρίζουμε ότι έχει κρίσιμο ρόλο να παίξει αυτό στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Θυμάμαι τη συζήτηση που κάναμε πριν από μερικές εβδομάδες. Τώρα είναι νέα η Επιτροπή μας, νέο το Κοινοβούλιο και φαίνεται αυτό, αλλά η ανησυχία παραμένει. Υπάρχει τεχνολογία, άραγε τι γίνεται. Τώρα θαύουμε διοξίδιο του άνθρακα. Αυτό είναι σαν να θαύουμε ραδιενεργά απόβλητα. Ας πούμε, μήπως πάθουμε τίποτα. Ε, όλες αυτές οι ερωτήσεις είναι ε, δεδομένες. Ε, όσο δαπανηρό και να είναι, ε, όσο χρησιμοποιούμε ακόμα ρηκτά καύσιμα, χρειάζεται αυτή η τεχνολογία. Και έχει σημασία να μην χασομερίσει η Ευρώπη και μας πάρουν άλλη τη σειρά και την πρωτοπορία σε αυτή τη τεχνολογία. Ελάτε λοιπόν στο σεμινάριο να μάθετε περισσότερα για το θέμα το μεσημέρι. Ευχαριστώ. <laughs> Πολύ κομψά τα λέτε. Για το πώς μπορεί κανείς να περάσει το μεσημεριανό του διάλειμμα. Στην Ουάσιγκτον μας είπανε ότι την Παρασκευή ξεκίνησε μια λειτουργία μια τέτοια μονάδα, η πρώτη μονάδα στη Βιρτζίνια. Δηλαδή και στι Ηνωμένε Πολιτείε υπάρχουν αυτά τα πράγματα και στην Κίνα και στην Ευρώπη. Και τίθεται το ερώτημα τι να κάνουμε το διοξίδιο του άνθρακα. Προφανώς πολύ σοβαρό θέμα και σημαντικό. Α, θα πρέπει λέει να κάνουμε τώρα δοκιμαστική ψηφοφορία, να δούμε αν λειτουργούν τα μηχανήματα. Λοιπόν, θα χιονίσει τα Χριστούγεννα, ναι ή όχι, αυτό ψηφίζουμε. <laughs> Τι πιστεύετε, όποιος θέλει να χιονίσει ε, πράσινο, όποιος δεν θέλει να χιονίσει κόκκινο και όποιος αδιαφορεί εποχή. Δοκιμαστική ψηφοφορία, θέλετε να χιονίσει τα Χριστούγεννα. Αλλά abgestimmt. Ψηφίσατε όλοι. Όχι. Fünf könnten auch abstimmen. Πέντε ακόμα περσεύουνε. Τι έγινε, δεν έχετε κάρτες. 55 είναι παρόντες. Okay. Ja, dann sagen wir mal Ende der Abstimmung. Καλά, ας πούμε λοιπόν πέρα στις ψηφοφορίες. Λοιπόν, ε, λοιπόν θα χιονίσει, λέει η συντριπτική πλειοψηφία. Ε, και λειτουργούν και τα μηχανήματα, ωραία. Super. Dann kommen wir... Ε, θαυμάσια. Συνεχίζουμε και περνάμε στην κανονική ψηφοφορία για την έκθεση της κυρίας Ρόσπα. Τροπολογία υπαριθμών 1. Ο κύριος Ταταρέλα, κάτι διαδικαστικό είχατε. Μικρό. μικρόφωνο. Η συζήτηση είναι ακόμα ανοιχτή. Ήθελα να παρέμβω για το θέμα. Σα ευχαριστώ Πρόεδρε. Ήθελα να υπογραμμίσω κάποια επιχειρήματα. Η ζωή στον πλανήτη Γη γεννήθηκε στην ε, θάλασσα κοντά σε πηγές ε, θιούχου υδρογόνου ε, υδραργύρου, συγγνώμη. Η Ιταλία έχει μια, καμιά δεκαριά τέτοιων ε, ε, μάλλον ηφαιστείων και ένα από τα πιο επικίνδυνα ηφαίστεια. Και τέτοιοι γίγαντες της φύσης μας έχουν δείξει πώς συμπεριφέρεται το διοξίδιο του άνθρακα στο υπέδαφος και πώς και αν μπορούμε να διαχειριστούμε τέτοιους κινδύνους. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε αυτές ε, τα επιστημονικά περίμετα που είναι στρατηγική σημασία για την εφαρμογή της ε, τεχνολογίας ε, αποθήκευσης και σύλληψης του διοξιδίου του άνθρακα για να μπορέσουμε να δούμε πώς αποθηκεύονται αυτά τα μεθάνιο, πώς μπορεί να αποθηκευτεί το μεθάνιο με ένα μεγάλο τμήμα της ενεργειακής επανάστασης θα γίνει γύρω από την καύση ορυκτών ε, καυσίμων και μέσω της σύλληψης και αποθήκευσης του διοξιδίου του άνθρακα. Όμως οι πολίτες μας γνωρίζουν πολύ λίγα όλα αυτά και θεωρώ πως αυτό είναι αδίκο και απαραδεκτό. Οι πληροφορίες είναι στρεβλωμένες υπέρ της ανανεώσιμης ενέργειας. Στην Ευρώπη δεν έχουμε χώρο και στις χώρες μας, οι χώρες μας είναι πολύ πυκνοκατοικημένες. Πιστεύετε πως για να αντικατασταθεί μια πυρηνική, ένας πυρηνικός αντιδραστήρας που καλύπτει κάποια εκτάρια θα ήταν ε, απαραίτητη απαραίτητα ε, πολλά πολλά εκτάρια στις ε, ακτές για τις ε, ανεμογεννήτριες ε, πράγμα το οποίο δεν είναι δυνατόν. Γι' αυτό θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι πρέπει να προωθηθούν όλες οι νέες ενεργειακές τεχνολογίες, τονίζοντας ιδιαίτερα το CSS που εφαρμόζεται όχι μόνο στις ε, ηλεκτροπαραγωγικές εγκαταστάσεις που βασίζονται στον άνθρακα, αλλά και σε, στα δηληστήρια, στα ναυπηγεία και ούτω καθεξής. Είναι ένα πλάνο τέτοιου τύπου απαραίτητο και οι επιχειρήσεις μας θα πρέπει να βρουν τα οικονομικά μέσα για να μειώσουν τα κόστη των εγκαταστάσεων σύλληψης και αποθήκευσης του διοξιδίου του άνθρακα. Σας ευχαριστώ. Κύριε Ταταρέλα, δεν ήθελα να σας διακόψω, αλλά η συζήτηση έχει τελειώσει. Είμαστε πλέον στην ψηφοφορία. Νομίζω θέλετε να πείτε τίποτα για την ε, ε, τροπολογία. Τη συζήτηση την κάναμε. Εντάξει, τα είπατε, τελειώσανε όμως αυτά. Δεν γίνεται τώρα συζήτηση, ψηφίζουμε. Ε, κυρία Ρόσπαχ, ξαναζήτησε το λόγο, παρακαλώ. Για την ψηφοφορία σας, παρακαλώ, τώρα μην μπούμε στην ουσία και στη διαμάχη. Ναι ή ναι, όχι, εντάξει. Θα ήθελα να ξεκαθίσω κάτι. Έχω την εντύπωση ότι ο κύριος Σαταρέλα πιστεύει ότι ε, τα αποθηκεύουμε στο βυθό. Όχι, στο πέδαφος, κάτω από το βυθό, στις, γεωλογικού στους γεωλογικούς σχηματισμούς. Θα ήθελα επίσης να ρωτήσω μήπως μπορούμε να ψηφίσουμε τις τέσσερις τροπολογίες on block. Μάλιστα. Αφού διευκρινίστηκε και αυτό μπορούμε να ψηφίσουμε. Η τροπολογία αριθμών 1 της κυρίας Ρόσπαχ ηλεκτρονικά ε, ψηφί υπέρ. Ε, Συγγνώμη, ζητάει ο πρόεδρος. Ε, αρχίζει η ψηφοφορία αφού είναι ηλεκτρονική. Ψηφίσατε όλοι πέρα. 50 υπέρ, 1 ε, κατά, μία αποχή εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία υπερθμών 4 του Κρήτον Αρσένη. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 49 υπέρ, 4 κατά εγκρίθηκε επίση, 2 της κυρίας Ρόσμπαχ. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 47 υπέρ, 4 κατά μία αποχή εγκρίνεται και η 3 της κυρίας Ρόσπαχ, αρχή ψηφοφορία. Πέρας. 47 υπέρ, 5 κατά μία αποχή επίσης εγκρίνεται. Ωραία. Πάμε στην τελική ψηφοφορία τώρα για την έκθεση αυτή. Αρχίζει. Η ψηφοφορία πέρας. 48 υπέρ. Ένας κατά τρεις αποχές. Συγχαρτήρια κυρία Ρόσβαχ, για την έκθεση αυτή. Ακολουθεί το σημείο 9 που λέει προφορική ερώτηση προς το Συμβούλιο για ένα περιβάλλον χωρίς καπνό. Το Συμβούλιο θέλει, λέει, την 1η Δεκεμβρίου να παρουσιάσει κάποια συμπεράσματα, να εγκρίνει μάλλον κάποια συμπεράσματα και το Κοινοβούλιο για λόγους χρονικούς περιορίζεται σε αυτού του είδους τη συμμετοχή. Είναι μόνο προφορική ερώτηση και οι πολιτικές ομάδες στο δεύτερο ψήφισμα, στη δεύτερη συγγνώμη ολομέλεια του Νοεμβρίου θα κάνουν Ψήφισμα. Η έδιτε Στρέλα έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Υπό την ιδιότητα μου της εισηγήτριας, τη συντάκτρια καλύτερα για αυτή τη γνωμοδότηση, ε, πρέπει να σας πω ότι είναι πάρα πολύ σκόπιμο να κάνουμε αυτή την προφορική ερώτηση προς το Συμβούλιο για τη δημιουργία χώρων χωρίς καπνό. το Συμβούλιο δεν περιμένει τη γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου. Αυτό είναι απαράδεκτο. Η σύσταση έφτασε στο Κοινοβούλιο, θυμίζω, το καλοκαίρι. Μετά τις ευρωεκλογέ δηλαδή και σε έκτακτες περιστάσεις ε, όπου είχαμε την αλλαγή των μελών του Κοινοβουλίου, τη συγκρότηση των επιτροπών σε σώμα, τις διάφορες αρμοδιότητες, ε, ανάληψη καθηκόντων των βουλευτών. Η δικιά μας επιτροπή εδώ περιβάλλοντος ε, συγκροτήθηκε σε σώμα το Σεπτέμβριο. Δηλαδή σε ένα μήνα και λιγότερο δεν μπορούσε να κάνει περισσότερη δουλειά από όσοι έκανε το Κοινοβούλιο. Και επειδή απαιτεί η διαδικασία λοιπόν μια σειρά συνεδριάσεων για να καταλήγουμε πάντα με συνένεση, έχουμε αυτές τις βαριές διαδικασίες. Κάνουμε συζητήσεις, ακούμε τους και συγητές, ε, ψηφίζουμε στην Επιτροπή, ζητούμε μεταφράσεις των κειμένων, μετά και άλλες συζητήσεις και στην Ολομέλεια η τελική ψηφοφορία για την έγκριση ή την απόρριψη. Λοιπόν, για λόγους χρονικούς ήταν αδύνατο εμείς να ανταποκριθούμε σε αυτά που μας ζητούσε το Συμβούλιο. Έτσι λοιπόν θεωρώ απαράδεκτη αυτή την τακτική. Αδιαφορεί το Συμβούλιο για τη γνώμη του Κοινοβουλίου. Και τελικά η Σουηδική Προεδρία, από ό,τι έχω καταλάβει, θέλει να ολοκληρώσει το θέμα αυτό πριν από το Δεκέμβριο. Το καταλαβαίνουμε αυτό, αλλά σας παρακαλώ, το καταλάβει και το Συμβούλιο τη δική μας θέση. Θέλουμε να γίνει συζήτηση από όλοι θεσμικά όργανα. Γι' αυτό και θίγουν αυτοί, κάνουν αυτή την ερώτηση οι συνάδελφοι, ώστε το Συμβούλιο να μας πει για ποιους λόγους θέλει να προχωρήσει χωρίς την ε, θέση του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ κύριε Στρέλα. Είπαμε ότι η συγκρότηση του Κοινοβουλίου σε σώμα ε, επίεσε τις διαδικασίες, δεν μπόρεσε το θέμα να ακολουθεί στην κανονική του πορεία στην Επιτροπή. Δεν βλέπω λοιπόν άλλα σχόλια ή παρατηρήσεις να θέλετε να κάνετε. Ας ψηφίσουμε αν θα πρέπει να γίνει αυτή η προφορική ερώτηση στο Συμβούλιο. Ηλεκτρονικά και πάλι αρχίζει τώρα η ψηφοφορία παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Αποτέλεσμα. 45 υπέρ, ένας ε, κατά, δύο αποχές. Εγκρίνεται λοιπόν η προφορική ερώτηση. Τώρα έχουμε μερικά λεπτά να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Στις 11 η ώρα ραντεβού με τον κύριο Δήμα. Μικρή διακοπή. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα συνεχίσουμε τη συνεδρίασή μας θα ήθελα να καλωσορίσω από την δεύτερη Βουλή του Ολλανδικού Κοινοβουλίου την κυρία Λίσπετ Σπίς που, της Επιτροπής Περιβάλλοντος εκεί. Σας καλωσορίζουμε. Πάντα χαιρόμαστε όταν έχουμε συναδέρφους από ε, τα Εθνικά Κοινοβούλια. Καλώς ήρθατε. Ε, εξίσου θα ήθελα να καλωσορίσω στην Επιτροπή μας τον Επίτροπο κύριο Δήμα. 33 μέρες μέχρι το ξεκίνημα της Διεθνούς Διάσκεψης για το Κλίμα στην Κοπενχάγη. Βλέπετε από ε, τους πολλούς παρόντες ε, πόσες προσδοκίες υπάρχουν για την διάσκεψη. Περιμένουμε αγωνίως ε, να ακούσουμε τι έχετε να μας πείτε για την κατάσταση των πραγμάτων, την προετοιμασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και όσον αφορά τη γέφυρα προς τους εταίρους μας στον κόσμο, τις Ηνωμένες Πολιτείες, ε, τις αναπτυσσόμενες χώρες κλπ. Να μην χάσουμε άλλο χρόνο. Σήμερα το πρωί είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση σχετικά με τον ε, κατάλογο διαρροής άνθρακα που έχετε υποβάλει για τη μετεκατάσταση των ε, επιχειρήσεων, των, των των εκπομπών ε, και θέλαμε να αναβάλουμε την συνέχεια της συζήτησης μέχρι να ακούσουμε τι έχετε να μας πείτε εσείς. Θέλουμε λοιπόν να μας πείτε το άρθρο 10β, πώς το ε, εφαρμόζει η Κομισιόν και πώς θα συμμετέχει το Κοινοβούλιο στην διαδικασία της συναπόφασης. Αυτά τα δύο θέματα συνδέονται στενά μεταξύ τους. Σας δίνω το λόγο, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε ε, απόψεις σχετικά με τις ιδέες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών με αντικείμενο το κλίμα η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Κοπενχάγη με έναρξη ε, στις 7 Δεκεμβρίου. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν ενεργό και είχαν ενεργό ρόλο στην προώθηση μιας φιλόδοξης ευρωπαϊκής πολιτικής σχετικά με το κλίμα, πρωτοστατώντας διεθνώς και κινητοποιώντας βασικούς εταίρους μεταξύ των αναπτυγμένων και αναπτυσσομένων χωρών. Και προσβλέπω στη συνέχιση ε, της στενής και καρποφόρας αυτής της συνεργασίας στην Κόπενχάγη και με ευχαρίστηση βλέπω ότι το Κοινοβούλιο θα ε, πάρει μέρος με σημαντική αντιπροσωπεία. Ας δούμε λοιπόν ποιες είναι οι κύριες προκλήσεις, τα κύρια προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε ώστε να καταλήξουμε σε συμφωνία στην Κοπενχάγη. Τρεις είναι οι κύριες προκλήσεις. Πρώτα-πρώτα με ποιο τρόπο θα εξασφαλιστεί ότι οι αναπτυγμένες χώρες θα υιοθετήσουν νομικά δεσμευτικούς στόχους μείωσης των εκπομπών επαρκώς τολμηρούς ώστε η υπερθέρμανση του πλανήτη να μην ξεπεράσει τους δύο βαθμούς Κελσίου. Δεύτερο, με ποιο τρόπο θα εξασφαλιστεί ότι οι, οι αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως οι μεγαλύτερες οικονομίες, θα λάβουν επαρκή μέτρα προετοιμα... Ε, περιορισμού του ρυθμού αύξησης των εκπομπών, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος τον οποίο ανέφερα προηγουμένως. Και τρίτο, με ποιο τρόπο θα διασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότησης ε, για τη στήριξη στις αναπτυσσόμενες χώρες ε, τόσο της αναγκαίας προσαρμογής προς τις κλιματικές αλλαγές, τις αλλαγές οι οποίες έχουν γίνει ήδη ε, και, τα, και τις επιπτώσεις και επίσης για τις ενέργειες εκείνες οι οποίες θα οδηγήσουν σε περιορισμό της εκπομπής ε, αερίων του θερμοκηπίου. Η διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα στην Κοπεχάγη θα αποτελέσει ορόσημο για τις διεθνείς προσπάθειες αντιμετώπισης κλιματικής αλλαγής. Τώρα είναι η στιγμή που εμείς η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρειαστεί να δώσουμε πρώτη το παράδειγμα. Οπωσδήποτε, όμως η Κοπενχάγη θα αποτελέσει ε, απλώς την αφετηρία μιας μίζωνος τροφής, η οποία ελπίζουμε και η οποία πρέπει να οδηγήσει τον κόσμο σε μια πορεία ε, οικονομίας χαμηλών εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα, χαμηλών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ήδη καταβάλει μεγάλη προσπάθεια. Ζητήσαμε επίμονα από τις αναπτυγμένες χώρες να πρωτοστατήσουν στη μείωση των εκπομπών ε, δεσμευόμενες συλλογικά να μειώσουν τις εκπομπές μέχρι το 2020 κατά 30% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 στο πλαίσιο μιας ισόρροπους ε, διεθνούς συμφωνίας. Φυσικά, οι στόχοι των επιμέρους χωρών θα πρέπει να αντανακλούν τις αντίστοιχες ικανότητες και μερίδια ευθύνης και στο πλαίσιο αυτό προτείναμε ένα ε, ισόρροπο συνδυασμό κριτηρίων όπως είναι τα εξής. Πρώτον, ικανότητα πληρωμής από τις χώρες, το, το πλούτο, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν ε, των χωρών, το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα, να είμαι πιο ακριβής. Δεύτερον, οι δυνατότητες μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις διάφορες χώρες. Τρίτον, ε, έγκαιρη εγχώρια δράση, ε, οι προσπάθειες τις οποίες έχουν κάνει οι χώρες μέχρι τώρα ε, για την μείωση των εκπομπών, πράγμα το οποίο έχει επιτευχθεί δηλαδή μέχρι τώρα ε, όλα τα προηγούμενα χρόνια και κυρίως μετά το 1990. Και ε, τέταρτο, το πώς αυξάνει ο πληθυσμός κάθε χώρας. Συνολικά αναμένω ότι τα κριτήρια που προτείνουμε θα οδηγήσουν σε ισόρροπη σειρά δεσμεύσεων από τις αναπτυγμένες χώρες με τον αντίστοιχο στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαμορφώνεται σε 30%. Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης τροφοδότησε σειρά πολυμερών και διμερών συζητήσεων με θετικά αποτελέσματα. Υπό την πίεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλες βιομηχανικές χώρες κατέθεσαν τις προτάσεις τους για δεσμεύσεις και ορισμένες βελτίωσαν και ε, ανύψωσαν το επίπεδο των φιλοδοξιών τους. Ιδίως ε, τελευταία η Ιαπωνία και η Αυστραλία. Βεβαίως, ορισμένες αναπτυγμένες χώρες χρειάζεται ακόμη να δεσμευθούν ακόμη περισσότερο ε, έτσι οι προσφορές ε, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ρωσίας, της Ουκρανίας και του Καναδά δεν είναι αρκετά φιλόδοξες. Τονίζουμε στους εταίρους μας από τις αναπτυγμένες χώρες ότι εάν δεν δράσουμε εμείς δεν μπορούμε να περιμένουμε από τις ταχαίως αναπτυσσόμενες οικονομίες να αναλάβουν εκείνες δράση στην κλίμακα που απαιτείται. Χρειάζεται όμως επίσης να είμαστε σαφείς στο ότι η ανάληψη δράσης από τις αναπτυσσόμενες χώρες, από τις αναπτυγμένες χώρες, από μόνη της δεν αρκεί. Οι εκτιμήσεις για την αύξηση των εκπομπών σε παγκόσμιο επίπεδο είναι σαφείς και κατηγορηματικές. και οι αναπτυσσόμενες χώρες, ιδιαίτερα οι μεγάλες οικονομίες, οι μεγάλες αναδυόμενες οικονομίες, πρέπει οπωσδήποτε να συμβάλλουν. Ε, δεν τους ζητάμε βεβαίως να υιοθετήσουν κατά το παρόν στάδιο απόλυτες μειώσεις των εκπομπών, ωστόσο θα χρειαστεί να επιβραδύνουν το ρυθμό αύξησης των εκπομπών τους, ώστε να τις συγκρατήσουν κατά 15 με 30% κάτω από τα επίπεδα που προβλέπονται για το 2020, εάν δεν ληφθούν μέτρα. Business as usual. Για να περιοριστεί η αύξηση της θερμοκρασίας στους δύο βαθμούς οι παγκόσμιες εκπομπές πρέπει να φτάσουν στο ανώτατο επίπεδό τους πριν από το 2020 και έπειτα να έχουν περιοριστεί μέχρι το 2050 τουλάχιστον κατά 50% έναντι των επιπέδων του 1990. Είναι απολύτως απαραίτητα οι, οι, οι, αναπτυγμένες χώρες να περιορίσουν την αύξηση των εκπομπών τους προκειμένου να επιτευχθούν οι ανωτέρω στόχοι. Στον Παλί τα μέλη της ε, ε, διάσκεψης συμφώνησαν ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες ε, θα λάβουν εθνικώς ενδεδειγμένα μέτρα μείωσης εκπομπών με τεχνολογική και χρηματοδοτική στηρίξη από τις αναπτυγμένες χώρες. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προτείνει οι αναπτυσσόμενες χώρες να καταρτήσουν εθνικά σχέδια οικονομικής ανάπτυξης με χαμηλά επίπεδα εκπομπών που θα περιλαμβάνουν δράσεις για τη μείωση των εκπομπών τους ε, στους κύριους τομείς της οικονομίας. Δηλαδή θα έχουν εθνικά σχέδια μείωσης των εκπομπών και τα εθνικά αυτά σχέδια θα περιέχουν συγκεκριμένες ενέργειες και πράξεις. Στα σχέδια αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνονται δράσεις οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν με εγχώριους πόρους μπορούν να υλοποιηθούν μέσω της αγοράς του διοξιδίου του άνθρακα, της παγκόσμιας αγοράς του διοξιδίου του άνθρακα και οι οποίες βασίζονται σε διεθνή χρηματοδοτική και τεχνολογική στήριξη που προέρχεται από τα δημόσια οικονομικά. Με βάση τα ανωτέρω σχέδια οικονομικής ανάπτυξης θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας συντονιστικός μηχανισμός ο οποίος θα ε, προχωρά σε εκτίμηση των αναγκών ε, που υπάρχουν και θα καταγράφει τις υφιστάμενες επιλογές για τη στήριξη της εφαρμογής των προγραμμάτων. Αποφασιστική σημασία είναι η χρηματοδοτική στήριξη από τις αναπτυγμένες χώρες των δράσεων των αναπτυσσόμενων χωρών για τη μείωση των εκπομπών τους. Η έλλειψη σημαντικής πρόοδος σήμερα στις διαπραγματεύσεις των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αδυναμία των αναπτυγμένων χωρών να προσφέρουν χρηματοδότηση. Το αδιέξοδο αυτό ακριβώς επιχειρήσαμε να άρουμε με την πρόσφατη ανακοίνωσή μας σχετικά με τη χρηματοδότηση των πολιτικών ε, ε, και των πολιτικών και των μέτρων για το κλίμα. Με βάση την απόφαση του τελευταίου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να προσφέρει το μερίδιο της χρηματοδότησης από δημόσιους πόρους που της αναλογεί. Το Συμβούλιο υιοθέτησε την εκτίμηση της Επιτροπής ότι θα απαιτηθούν ε, περίπου 100 δισεκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση ως το 2020 προκειμένου να καλυφθεί το οριακό κόστος των μέτρων για το κλίμα στις αναπτυσσόμενες χώρες, το επιπρόσθετο κόστος. Το κόστος αυτό θα καλυφθεί μέσω ενός συνδυασμού εθνικών μέτρων των χωρών αυτών, της αγοράς του διοξιδίου του άνθρακα εκπομπών και της ε, διεθνούς δημόσιας χρηματοδότησης. Το συνολικό ύψος της απαιτούμενης διεθνούς χρηματοδότησης ε, εκτιμάται ότι θα κυμαίνεται μεταξύ 22 και 50 δισεκατομμυρίων ευρώ σε αιτήσια βάση από το 2020. Εάν το ποσό αυτό επιμεριστεί και ληφθεί υπόψη η χρηματοδοτική ικανότητα των χωρών, η ευθύνη για τις εκπομπές, καθώς και η συνεισφορά των ταχαίως αναπτυσσομένων χωρών ε, τότε το μερίδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ανέλθει από 2 15 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως ε, το 2020. Αυτό ίσως θα μπορέσω να το εξηγήσω στη συνέχεια αν ερωτηθώ. Για την περίοδο μετά το 2013 η Επιτροπή θα καταρτήσει πρόταση για ενιαία συνολική προσφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξετάζοντας το ενδεχόμενα χρησιμοποίηση του κοινοτικού προϋπολογισμού, μια περίπτωση η οποία επιτρέπει και την ε, εμπλοκή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά επίσης και την ιδέα ενός ταμείου κλίματος ε, και τον τρόπο με τον οποίο άμεσες συνεισφορές από τα κράτη-μέλη μπορούν να συμβάλλουν εντασσόμενες στη συνολική κοινωτική προσπάθεια. Όπως όμως ε, παραδέχθηκε και το Ευρωπαϊκό Συμβουλίο, υπάρχει και τώρα ανάγκη χρηματοδοτικής στήριξης και όχι μόνο μετά το 2013. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο ε, για το διάστημα 2010-2013 η Επιτροπή πρότεινε έγκαιρη χρηματοδότηση προς τις αναπτυσσόμενες χώρες της τάξης των 5 7 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Βασιζόμαστε στην υποστήριξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ε, ε, διάδοση και προώθηση των τολμηρών επιδιώξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το κλίμα, τις διάφορες επαφές σας, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές με συναδέλφους σας των άλλων κοινοβουλίων ανά τον κόσμο, και ξέρω ότι ήσασταν πρόσφατα την περασμένη εβδομάδα στις Ηνωμένε Πολιτείε και είχατε σημαντικές επαφές με μέλη του Κογκρέσου και θα είναι ενδιαφέρον να μάθουμε περισσότερα για αυτές τις επαφές ε, και βεβαίως με τους επιχειρηματικούς κύκλους και με την ευρύτερη κοινωνία των πολιτών. Ε, και θέλω να σας ευχαριστήσω για τις προσπάθειες που καταβάλατε ε, ε όλον αυτόν τον καιρό ε, και για την εξαιρετική συνεργασία την οποία είχαμε ε, συνεχώς. Επίσης θα ήθελα να χαιρετήσω την πρωτοβουλία σας για τη διατύπωση ψηφίσματος προς έκδοση ε, αργότερα εντός του μηνός σχετικά με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Διάσκεψη Κοπεχάγης. Ειδικότερα συμμερίζομαι την έκκληση του Κοινοβουλίου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να αγωνιστεί για την επίτευξη συμφωνίας στην Κοπενχάγη, η οποία θα συνάδει με τον στόχο των δύο βαθμών αύξησης της θερμοκρασίας για τον οποίο απαιτούνται δραστικά μέτρα εκ μέρους τόσο των αναπτυγμένων όσο και των αναπτυσσόμενων χωρών. Στο πλαίσιο αυτό η Επιτροπή διαπιστώνει με ικανοποίηση ε, στο σχέδιο ψηφίσματος του Κοινοβουλίου την ένθερμη υποστήριξη ε, ε, λύσεων που βασίζονται στην αγορά και του αναμορφωμένου μηχανισμού καθαρής ανάπτυξης σε μια μελλοντική συμφωνία όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών που οφείλονται στην ε, ε, αποδάσωση και την υποβάθμιση των δασών, η Επιτροπή επιθυμεί να επαναδιακηρύξει ότι πράγματι θα αγωνιστεί για την πρόθεση αυστηρών κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων και ότι θα συνεκτιμήσει τις επιπτώσεις στη βιοπικιλότητα. Γιατί μπορεί να ε, συμφωνούμε όλοι ότι οι κλιματικές αλλαγές είναι παγκόσμιο απειλή την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε και μάλιστα επειδή του χρόνου θα είναι και το παγκόσμιο έτος βιοπικιλότητας, ότι η άλλη μεγάλη και άμεσα συνδεόμενη με τις κλιματικές αλλαγές απειλή για τον πλανήτη είναι η απώλεια της βιοπικιλότητας. Ε, perhaps I'll carry on possible questions regarding the issue, or shall I just make a statement? Okay. Just do it now. Okay. Um, regarding uh, uh, this, Όσον αφορά την απόφαση αυτή που αφορά τους τομείς ε, που είναι πιθανό να ε, υπόκεινται σε διαρροή άνθρακα κατάσταση των εκπομπών. Σημαντικό είναι να τονίσουμε ότι η απόφαση αυτή ε, σχετίζεται με το μονομερές σενάριο της μείωσης των 20% σε περίπτωση ε, που, οι άλλες χώρες δεν θα ε, αναλάβουν υποχρεώσεις για μείωση των εκπομπών και θα αναθεωρηθεί το 2014 με βάση τα αποτελέσματα της Κοπεχάγης. Μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2010 η Κομισιόν βάσει τα αποτελέσματα των διεθνών διαπραγματεύσεων θα υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θα ε, θα υποβάλει στο Κοινοβούλιο πρόταση που θα συνοδεύεται από σχετικέ προτάσει. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα επιβεβαίωσε ότι ο κατάλογο θα αναθεωρηθεί υπό το φω των αποτελεσμάτων ε, των διεθνών διαπραγματεύσεων για την αλλαγή του κλίματο. Παραθέτω απευθεία από την παράγραφο 22 των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Οποιαδήποτε τέτοια πρόταση θα αποτελεί σε αντικείμενο απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και όχι της διαδικασίας της επιτροπολογίας. Όσον αφορά την ψηφοφορία σας για την απόφαση που αφορά τους τομείς ε, που ε, θεωρείται πιθανό να αποτελέσουν αντικείμενο διαρροής άνθρακα. Πιστεύω ότι η απόφαση αυτή νομικά στέκει και να σας εξηγήσω γιατί το άρθρο 10α αναφέρει ότι ο κατάλογος που αναφέρεται στην παράγραφο 13 θα συντάσσεται έχοντας λάβει υπόψη τα, τα υπάρχοντα στοιχεία, τα στοιχεία που διατίθενται. Χώρες που αποτελούν ε, χώρες που αντιπροσωπεύουν σημαντικό μέρος ε, της ε, διεθνούς ε, παραγωγής, καθώς και χώρες που έχουν αναλάβει διεθνείς υποχρεώσεις σχετικά με την μειωσή των εκπομπών. Σε περίπτωση που οι εκπομπές των χωρών αυτών είναι συγκρίσιμες με τις Ευρωπαϊκή Ένωσης, η ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει λάβει υπόψη και τα δύο αυτά κριτήρια στο, στην αιτιολογική σκέψη 22. Στην παρούσα φάση μόνο η Νορβηγία, η Ισλανδία και η Ελβετία έχουν δεσμευτεί να μειώσουν τις εκπομπές ε, στους σχετικούς τομείς. Οι χώρες αυτές μαζί δεν αντιπροσωπεύουν σημαντικό μερίδιο της ε, παγκόσμιας παραγωγής σε τομείς που θεωρείται ότι κινδυνεύουν να αποτελέσουν αντικείμενο διαρροής άνθρακα. Επίσης ε, δεν υπάρχουν ε, ε, διαθέσιμα στοιχεία λόγω της μη συγκρισιμότητα των στοιχείων και της έλλειψη διεθνών στοιχείων ανατομέα καθότι το σχέδιο απόφασης ε, αναφέρει ότι μόνο η Νορβηγία, η Ισλανδία και Ελβετία ε, έχουν δεσμευτεί να μειώσουν τις εκπομπές και δεν αντιπροσωπεύουν σημαντικό μερίδιο της διεθνούς παραγωγής, δεν έχει νόημα και δεν ε, θεωρείται απαραίτητο να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητά τους ως προς τις εκπομπές. Επειδή κάποιες χώρες μπορεί να διαφωνήσουν με κάτι τέτοιο, η Κομισιόν προχώρησε ένα βήμα πιο πέρα. Έγινε μια μελέτη για την Επιτροπή που έχει να κάνει με την αποτελεσματικότητα άνθρακα παγκοσμίω με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία. Ε, κατά τη γνώμη της Επιτροπής τα στοιχεία αυτά δεν είναι ε, αρκετά αξιόπιστα ώστε να ληφθούν υπόψη. Η μελέτη αυτή θα δημοσιευτεί από την Επιτροπή. Τέλος, η Επιτροπή Περιβάλλοντος ε, στο στην πρόταση ψηφίσματο για συμπεράσματα τη Κοπεχάγη δηλώνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η μόνη, ο μόνο περιφερειακό φορέα στον κόσμο που έχει αναλάβει δεσμευτικού στόχου για την μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, υιοθετώντα ε, το σχετικό κλιματικό πακέτο. η Κομισιόν ε, περιμένει από τρίτες χώρες ε, να αναλάβουν υποχρεώσεις για μείωση των ε, εκπομπών. Η απόφαση που αφορά τους τομείς που μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο μετακατάστασης των εκπομπών αντικατοπτρίζει την κατάσταση πριν την Κοπεχάγη θα αναθεωρηθεί υπό το φως των αποτελεσμάτων της Κοπεχάγης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε ε, για την παρουσίαση αυτή. Σαφής η ε, ρίση. Μετά την Κοπεχάγη θα αναθεωρηθεί ο κατάλογος με συμμετοχή του Κοινοβουλίου. Άλλωστε το λέει και η νομοθεσία αυτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, φαντάζομαι ότι θέλετε να πείτε όλοι κάτι, να μιλήσετε όλοι. Δυστυχώς δεν προλαβαίνουμε όλοι. 26 συνάδελφοι ζήτησαν το λόγο, 27. Κλείνει ο κατάλογος τώρα, έκλεισε. 27 συνάδελφοι. Ε, δεν χωράει. Λυπάμαι πάρα πολύ. 1,5 λεπτό ο καθένας, θα κάνω ό,τι μπορώ και θα είμαι και αυστηρός. Αλλιώς είναι άδικο απέναντι σε εκείνους που δεν θα πάρουν το λόγο. Λοιπόν, πρώτος ο Καρχάινς Φλόρεντς, 1,5 λεπτό από τώρα. Θα προσπαθήσω σύντομα. Ε, και ή δυνατόν ερωτήσεις για την Κοπεχάγη όχι γενικές φιλοσοφικές τοποθετήσεις. Ε, και αυτό ισχύει για όλους, όχι μόνο για το Florence. Υποθέτω ότι αυτό το αφαιρείται από το χρόνο μου, έτσι. Αλλιώς έχω ακόμα λιγότερο χρόνο. Κύριε Επίτροπε, αναφερθήκατε στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την περιγράψατε. Αλλά ποια είναι η διαπραγματευτική στρατηγική. Ποια είναι η στάση και η δράση. 31 ημέρες ε, είναι μέχρι την Κοπεχάγη και είναι πολύ χρόνος αυτός βλέπετε ελπιδοφόρα μηνύματα και ποια είναι τα προβλήματα και δυσκολίες. Και δεύτερη ερώτηση. Ε, χτες το βράδυ, από ό,τι φαίνεται, ε, υπήρξε αντιπροσωπεία ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών υπό την αιγησία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρουσία εκπροσώπων του Συμβουλίου. Ποια είναι η διαπραγματευτική στρατηγική που προέκυψε. Η Λίντα Μακάβαν. Σα ευχαριστώ πολύ σύντομα, Επίτροπε. Την περασμένη εβδομάδα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συζητήθηκαν τα οικονομικά, αλλά δεν δόθηκαν ε, στοιχεία αριθμητικά για το πόσο θα χρηματοδοθεί. Λοιπόν, πόσο μεγάλο μπορεί να είναι αυτό το πρόβλημα στι διεθνεί διαπραγματεύσει επειδή η Ευρώπη θέλει να ηγηθεί και έπειτα για το θέμα τη διαρροή του άνθρακα που, είπατε, που θα το ψηφίσουμε. Είπατε ότι οι διεθνεί ε, θα προσπαθήσουν να μειώσουν το διοξίδιο του άνθρακα που εκπέμπουν και θα δεσμευτούν γι' αυτό. Αν ας πούμε αν είπα φτιάξουν ένα σύστημα συγκρίσιμο με το δικό μας, αυτό θα σημαίνει μάνι, ότι κάποιοι από τους τομείς που έχετε εδώ εντοπίσει στη λίστα θα μπορούσαν να βγουν από τη λίστα. Και αυτή η λίστα, ό,τι μορφή και αν πάρει θα επανέλθει ε, στη διαδικασία συναπόφασης με βάση το 10β. Ευχαριστώ, Chris Davis. Πρόεδρε, ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να ξανακούσουμε τον Επίτροπο, αλλά εάν όχι, θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία για να τον ευχαριστήσω και αυτόν και την ομάδα του για το έργο του κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών. Ξέρω πως ε, περάσαν πολλά δύσκολα και πράγματα και επικρίσεις ακούστηκαν, αλλά για την ατζέντα για τις κλιματικές αλλαγές μας έχει κάνει όλους περήφανους. Σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Να πω τώρα δύο πράγματα για την Κοπενχάγη. Πριν από δύο ε, μήνες ο Αντρέα Γκόλγαν μας είπε ότι ο ελάχιστο στόχος για να κρίνει ένα επιτυχές αποτέλεσμα θα ήταν το να συμφωνήσουμε ότι δημιουργήθηκαν μέτρα για να μην αυξηθούν πάνω από δύο αυξηθεί η θερμοκρασία πάνω από δύο βαθμού, ότι θα συμμετέχουν όλες οι πιο μεγάλες χώρε και ότι θα μπορούσε να βελτιώνεται και να με βάση τις εξελίξεις, τις γνώσεις κτλ. Τώρα ακούσαμε πως ε, αυτοί οι στόχοι έχουν κάπως αυληθεί από τη ΑΕΠΑ, από τι προσπαθούμε να φτιάξουμε, μια πολιτική δομή, ώστε μια μελλοντική διάσκεψη να διασφαλίσει ε, ε, ε, συμφωνία. Μπορείτε να μας εξηγήσετε τι σημαίνει αυτό, ποια είναι τα ελάχιστα προποτήματα για να θεωρήσετε ότι επιτύχατε θα το χάσει. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον Επίτροπο που ήρθε εδώ. Μια ερώτηση που σχετίζεται με αυτό την υπόθεση της διαρροή του άνθρακα. Είπατε πως ο κατάλογος που έχουμε σήμερα μπροστά μα ισχύει για το μονο, τη μονομερή μείωση του 20%. Βασίζεται στην υπόθεση ότι κανείς άλλος εκτός της Ένωσης δεν ε, κάνει κάτι σχετικά με αυτή την υπόθεση. Όμως, ποια είναι η εκτίμησή σα επειδή ήσασταν στι διαπραγματεύσει, ποια είναι η πραγματική κατάσταση το, όσον αφορά τις δεσμεύσεις ε, των άλλων χωρών. Θεωρείτε πως ε, κανένας άλλος δεν κάνει τίποτα ή ότι και άλλοι μεγάλοι παίχτες προσπαθούν. Ποια είναι η δική σας αξιολόγηση για την πραγματική κατάσταση και είπατε ότι ο κατάλογος για τη διαρροή του άνθρακα θα αναφερθεί μετά από την Κοπενχάγη και αυτό θα γίνει με τη συναπόφαση. Εσείς τι φαντάζεστε, πιστεύετε πραγματικά ότι στην συναπόφαση, στη διαδικασία συναπόφασης μετά από την Κοπενχάγη σε κάθε τομέα, μάλλον οποιοδήποτε τομέα θα βγει πραγματικά από τον κατάλογο. Δεν φοβάστε πως όλες αυτές οι ομάδες πίεσης θα πούν που αυτό είναι ένα όφελος που έχουμε επιτύχει, άρα θα το διατηρήσουμε. Thank you. Ε, Ευχαριστώ, Μύρος Λαφούτσκι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καλώς ορίσατε, κύριε Επίτροπε. Χαίρομαι που σας βλέπω. παραμονές της ε, διάσκεψης της Κοπενχάγης. Έχω την εξή ερώτηση. Όταν συζητάμε για διαπραγματεύσεις στην παγκοσμιοποίηση, ε, ζητούμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιαπωνία και την Κίνα. Προσωπικά πιστεύω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα θα είναι η Ινδία. Έχετε εσείς καμία πληροφόρηση για τη τρέχουσα θέση της Ινδίας, ε, που είναι μια οικονομία που αναπτύσσεται με πολύ γοργούς ρυθμούς. Και όταν μιλάμε για ρήπανση, νομίζω ότι είναι η τρίτη στον κόσμο από πλευρά ε, ρήπανση. Ευχαριστώ, κύριο Ρώση. Ευχαριστώ. Ε, Επίτροπε Δήμα, εγώ είμαι απογοητευμένο από την δική σα παρέμβαση. Περίμενα ότι από έναν τόσο έμπειρο πολιτικό θα είχαμε περισσότερη στήριξη. Μιλήσατε για τρει στόχου. Μείωση των εκπομπών στι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, κόστο για την βιομηχανία, εγγυήσει για τι αναπτυσσόμενες χώρε που περιορίζουν τι εκπομπέ του, αλλά αυτό συνδέεται με χρηματοδότηση που πληρώνουν οι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση για να στηριχθούν οι αναπτυσσόμενε χώρε ακριβώ. Άρα δηλαδή για να στηρίξουμε τεχνολογική καινοτομία, αυτών των βιομηχανιών που είναι ανταγωνιστικέ των δικών μα. Δηλαδή, ο στόχο σα είναι να χρηματοδοτήσετε ε, βιομηχανίε των τρίτων χωρών για να βελτιώσουν τι τεχνολογίε του, για να μα κάνουν καλύτερο ανταγωνισμό στι δικέ μα, να υποχρεώσετε τι δικέ μα ε, επιχειρήσει σε περισσότερου περιορισμού των εκπομπών. Αν αυτή είναι η στόχη που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εγώ ω Ευρωπαίο πραγματικά έχω τρομοκρατηθεί για το ποιοι θα ζημιωθούν από την μετεγκατάσταση των βιομηχανιών μα από την Ευρώπη στι τρίτε χώρε. Ε, από εδώ μόνο κόστη, από εκεί μόνο συμβολές για να βελτιωθεί η τεχνολογία. Εγώ πιστεύω πως η Ευρωπαϊκή Κομισιόν θα πρέπει να κάνει μια πολύ σοβαρή αυτοκριτική. εγώ περίμενα από εσά να ακούσω παρηγορητικά λόγια, λόγια παρηγοριάς για τις επιχειρήσεις που περνούν κρίση στην Ευρώπη. Όχι χρηματοδότηση των ε, ανταγωνιστών τους και παραπάνω δαπάνες για τις δικές μας επιχειρήσεις. Ευχαριστώ. Ρίχα Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να, με λίγα δευτερόλεπτα να τα αφιερώσω σε ευχαριστίες στον Επίτροπο για το έργο του υπέρ του περιβάλλοντος και πώς σκέφτεται να συμπελάβει στη διαπραγματευτική ομάδα την αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γιατί συνήθω στο περιθώριο καθόμαστε. Θα πάνε πολλοί συνάδελφοι στην Κοπεχάγη. Εσείς πώς θέλετε να μας ε, συμπεριλάβετε στις εργασίες σας, γιατί είμαστε και ο ημάντας μεταβίβασης προς τους ε, Ευρωπαίους πολίτες που μας εξέλεξαν. Γίνεται μεγάλος λόγος για την Κίνα, την Ιαπωνία ε, και τις ε, Ηνωμένε Πολιτείες στην ενεργειακή απόδοση και όχι τη μείωση του διοξιδίου του άνθρακα. Είναι θετική λοιπόν αυτή η πορεία σε σχέση με την Κοπεχάγη ή αρνητική. Και το πρόβλημα της οικονομίας είναι ότι με το σύστημα ETS ε, εμπορίας εκπομπών χάνονται σημαντικοί πόροι που κανονικά θα πήγαιναν σε απαραίτητες επενδύσεις. Σε άλλα μέρη της γης αυτό δεν συμβαίνει. Πώς μπορούμε να βεβαιωθούμε ότι ε, τα χρήματα θα παραμείνουν στις επιχειρήσεις για να μπορέσουν να κάνουν τις επενδύσεις που χρειάζονται. Γιατί είναι σκληρός ο παγκόσμιος ανταγωνισμός. Ευχαριστώ. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Και εγώ, όπως οι συνάδελφοι τον κύριο Επίτροπο, παραμονές της Κοπενχάγης και στην προετοιμασία της, δεν άκουσα πολλά για το ρόλο που ε, θα μπορούσε να διαδραματίσει το πολύ σοβαρό το δάσος στην καταπολέμηση κλιματικής αλλαγής. Θα ήθελα την αίσθησή σας, γιατί μιλάμε για την αποψήλωση και την καταπολέμησή της, αλλά πολύ συχνά ξεχνάμε την προώθηση της αηφόρου δασοκομείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και νομίζω ότι θα πρέπει να ε, υπογραμμιστεί και αυτό. Σε ό,τι αφορά την αποψήλωση των δασών, ακόμα και αν το θέμα διεθνούς συμφωνίας για τη χρηματοδότηση ε, παραμένει η καρδιά του προβλήματος, υπάρχει και ένα ζήτημα ευαισθητοποίησης των ε, τροπικών κρατών για τον έλεγχο και εφαρμογή εθνικών προγραμμάτων κατά της αποψήλωσης των δασών. Και αξίζει ε, να τονιστεί. Στα πλαίσια της πρωτοβουλίας RED, για παράδειγμα, τι θα κάνουμε πώς μπορούν οι βιομηχανικές χώρες να ζητήσουν από τις αναπτυσσόμενες κάποιες δεσμεύσεις. Τι προτίθεται να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βεβαιωθεί ότι οι χώρες αυτές θα συμμετέχουν πλήρως στα προγράμματα ε, συνεργασίας κατά της αποψήλωσης των δασών. Επιπλέον, εκτός από αυτά τα μέτρα εξωτερικής συνεργασίας για την καταπολέμηση της αποψήλωσης, Μερσή, διακόπτει ο Πρόεδρος, τελείωσε ο χρόνος σας. Ε, ε, σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Δήμα, εγώ σας ευχαριστώ για τη μεγάλη προσοχή που δώσατε στο συναγερμό των πολιτών της ε, Μεσογείου για τα τοξικά απόβλητα ε, εκεί. Υπάρχουν κάποιες διαρροές εκεί και δώσατε μεγάλη προσοχή σε αυτή την υπόθεση. Και έπειτα με μεγάλη προσοχή παρακολούθησα την παρέμβασή σας ε, με την οποία θίξατε διάφορα μεγάλα προβλήματα της Ευρώπης που βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη της Ευρώπης, της ίδιας και της Κομισιόν, αλλά και επαναλαμβάνω συζητώνται και εδώ στην Επιτροπή μας. Εγώ πιστεύω πως ε, η παράβασή σας ήταν ε, πολύ πλήρης ε, και σύμφωνα με τα ερωτήματα που σας απευθύνθηκαν θα μας δώσετε και πιο συγκεκριμένες ιδέες για το πώς θα προχωρήσουμε. Όμως το πιο πολύ, αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο και ολοκληρώνω είναι ότι μετά από την Κοπεχάγη σίγουρα θα έχουμε τρόπο να συζητήσουμε τα αποτελέσματα αυτής της διάσκεψης εδώ στην Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μα για την προστασία του κλίματος συζητάμε τώρα τα αναβάγια με τα τοξικά απόβλητα στη Μεσόγειο. Αν θέλετε μπορείτε να απαντήσετε. Ο Κρήτον Αρσένης παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, είναι πάλι χαρά μας να σας έχουμε εδώ πέρα. Ε, στη τελευταία διάσκεψη, στη διάσκεψη των μερών στην Μπαγκόγκο, διαπραγματευτή τη Ευρωπαϊκή Ένωση αποχώρησε από την ε, COP15 και τάχθηκε υπέρ μια νέα συνθήκη σε συμφωνία με τη ΣΥΠΑ. Όμω, κατά τι επαφέ τη αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου στην Ουάσιγκτον με μέλη του Κογκρέσου, κατέστησε σαφέ ότι θα είναι πολύ δύσκολο για τη ΣΥΠΑ να επικυριώσουν οποιαδήποτε συμφωνία, καθώ κάτι τέτοιο απαιτεί 67 ψήφου από τι 100 τη γερουσία των ΗΠΑ. Ήδη 60 ψήφοι για την νομοθεσία που πετούνται στη Γερουσία είναι πάρα πολύ δύσκολοι να βρεθούν. Μήπω θα πρέπει λοιπόν να επαναξεταστεί η στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση για πραγματεύσει, καθώ φαίνεται ότι η ΗΠΑ ναι, με διατίθεται να περιορίσουν τι εκπομπέ, αλλά όχι να συμμετέχουν σε μια διεθνή δεσμευτική συμφωνία με ποσοτικού και μετρήσιμου στόχου. Ε, από την άλλη, σε αντίθεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ΗΠΑ έχουν ψηφίσει στην Βουλή των Αντιπροσώπων ήδη περίπου 5 δι για την προστασία των δασών του κόσμου προτίθεται η Ευρωπαϊκή Ένωση προς αυτήν την κατεύθυνση να πάρει συγκεκριμένα δεσμευτικά ποσοτικά αντίστοιχα μέτρα. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ. Ο κύριος Παναγιώτοφ. Παναγιώτοφ. Thank you. Σας ευχαριστώ. Εγώ θέλω να πω αν ευχαριστώ για την αντιπροσωπεία Μάλλον θέλω να σας ενημερώσω για την αντιπροσωπεία στην Washington. Δύο λόγια μόνο για να σας ενημερώσω. Ήταν μια αντιπροσωπεία που μετέβη στην Ουάσιγκτον πέντε βουλευτές με τον κύριο Τζο Λάινεν. Πολύ δύσκολη και σκληρή συζήτηση, αλλά τελικά είμαι πεπισμένος πως ο πάγος λιώνει ε, η βασική συμβολή ήταν του κυρίου Τζο Λάινερ γιατί τους έπεισε σε μια πολύ δύσκολη συνέντευξη τύπου πως όλα αυτά είναι πολύ χρήσιμα και πολύ επωφελή για όλους ε, γιατί είναι πολύ πρακτικά τα θέματα έδωξε μεγάλη αντοχή σε πολύ δύσκολες συζητήσεις και γι' αυτό πιστεύω πως είναι απαραίτητο αυτός ο διάλογος να γίνεται όλο και πιο εντατικά ώστε να ε, είναι επιτυχής. Σας ευχαριστώ. Ε, Σας ευχαριστώ για τα λουλούδια αυτά. Θα ήταν ε, υπερβολικό ε, εάν ε, οι συνεντεύξει τύπου μας άλλαζαν τη γνώμη της Αμερικανικής Γερουσίας, αλλά μπορεί να συμβάλαμε κάπως ε, στην πρόοδο. Υπάρχουν άλλοι αποφασιστικοί παράγοντες. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φαντάλν. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, καλώς ορίσατε σας υποστηρίζουμε για την Κοπεχάγη σημαντικά θέματα. Σωστά αναφερθήκατε στη βιοπικιλότητα και στην αποψήλωση των δασών. Και ακριβώς αυτό το δεύτερο έχω συγκεκριμένη ερώτηση να σας απευθύνω. Την εξή. Για την καταπολέμηση της αποψήλωσης περιμένουμε πολλά από την αγορά. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα ε, με τα αγγλικά ίσως, σε περισσότερες γλώσσες. Γερμανικά έχουμε. Ελληνικά έχουμε. Αγγλικά έχουμε. Τώρα έχουμε και αγγλικά. Ελληνικά έχουμε. Ιταλικά. Ωραία. Από ό,τι φαίνεται λειτουργεί τώρα η διερμηνία. Μικρόφωνο δεν έχουμε τώρα. έλεγα λοιπόν... Ε, εντάξει ότι σωστά αναφερθήκατε ε, στην αποψήλωση των δασών και έχω συγκεκριμένη ερώτηση θα πρέπει ε, να δούμε ποια είναι ε, η αγορά αυτή, το κόστος, ε, οι κίνδυνοι που συνδέονται. Απέχουμε ακόμα από το στόχο το 2020 που είπαμε μείωση στο 50% πώς προχωρούμε σε αυτή την προσπάθεια, πώς μπορούμε να περιορίσουμε την αποψήλωση των δασών μέχρι τότε. Ευχαριστώ. Ο Μπάς Εκχάουτ. Yes, I'm also not talking about the flowers, but talking about ε, δεν θα μιλήσω για λουλούδια, για τα βάση. Μια πολύ σύντομη και συγκεκριμένη ερώτηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπέρ του να επιτρέψει βιομηχανικές χώρες να χρησιμοποιούν, να χρησιμοποιούν το, τις κόκκινες πιστώσεις μέχρι το 2020 ε, και πώς μπορεί να γίνει αυτό χωρίς ε, να υπονομεύσουμε την ε, περιβαλλοντική αποτελεσματικότητα των μειώσεων στο παράρτημα 1. Και για την Μπαγκόκ αναφέρθηκαν τα χέγγια για να αποφύγουμε τα φυσικά δάση να γίνουν φυτίες δασών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν υπέρ στην Μπαγκόκ, αλλά είπε αργότερα ότι είναι λάθος. Ελπίζουμε λοιπόν στη Βαρκελόνη τα, τα, σημεία αυτά που αφορούσαν τα δάση να επανέλθουν στο κείμενο. Μέχρι στιγμής όμως δεν έχουν συμπεριληφθεί πάλι στο κείμενο. Παρακαλώ λοιπόν τον Επίτροπο να μου ξεκαθαρίσει ότι θα συμπεριληφθούν πάλι τα κείμενα αυτά στη συμφωνία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πίτερ Λίζε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και εγώ τον Επίτροπο κύριο Δήμα για την καλή συνεργασία που είχαμε τα τελευταία χρόνια. Πιστεύω και θέλω να το πω αυτό προσωπικά ε, στον Επίτροπο. Όσον αφορά τη διαρροή άνθρακα έχετε κάνει πολύ καλή δουλειά. Και έχετε κάνει πολύ καλή προκαταρκτική δουλειά όσον αφορά τη χρηματοδότηση. Αναφέρετε στο ε, ε, έγγραφό σας την αρμοδιότητα του Κοινοβουλίου όσον αφορά τον προϋπολογισμό. Θα πρέπει να το έχουμε αυτό κατά νου, διότι όταν δίνουμε εκατομμύρια ευρώ θα πρέπει να συναποφασίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ώστε να φροντίσουμε να συμβάλλουν οι δαπάνες αυτές ε, στην καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος. Θα ήθελα να ρωτήσω, υπό ποιε συνθήκε, υπό ποιε προποθέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διατεθειμένη να περάσει από το 20% στο 30%, τι θα πρέπει δηλαδή να έχουμε από τις τρίτες χώρε και επίσης όσον αφορά τις αερομεταφορές και τις θαλάσσιες μεταφορές. Στους τομείς αυτούς ε, δεν είναι πολύ φιλόδοξο το κείμενο, ε, το, η Σύνδεση Κορυφή δεν είπε τίποτα για αυτό. Ε, έχουμε ένα νέο αποδυναμωμένο στόχο όσον αφορά τι αερομεταφορές. Το χειρότερο θεωρώ είναι ότι κύριε πίτροπε στην τελευταία ολομέλεια όπου ψηφίσαμε για τις, όπου μιλήσατε για τις αερομεταφορές, μας είπατε ότι ο πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή. Όχι, πρέπει να θέσω την ερώτηση, λέει ο κύριε Λίζε. Κύριε ε, Επίτροπε, έχει καθυστερήσει η σχετική πρόταση. Θα μπορούσατε να τα πείτε αυτά και πιο σύντομα. Κυρία Φρανσουά Κροστέτ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να επανέλθω στο θέμα της διαρροής ε, του διοξιδίου του άνθρακα. Βεβαίως θα πρέπει να ε, τηρήσουμε τις δεσμεύσει μας, αλλά οι διεθνείς συμβάσεις δεν κάνουν διάκριση μεταξύ των αναπτυσσομένων κρατών και δεν λαμβάνουν υπόψη τις πιο προηγμένες αναπτυσσόμενες χώρες. Βλέπε Κίνα. Η ε, οικονομική της ανάπτυξη ε, τρέχει και καλά κάνει. Αλλά η Ινδία, Κίνα, Βραζιλία δεν μπορούν να θεωρούνται, δεν θεωρούνται χώρες που θα πρέπει όσο και εμείς να μειώνουν ε, τα αέρια του θερμοκηπίου, ενώ είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής άνθρακα και παραγωγής διοξιδίου. Λοιπόν, εσείς τι λέτε γι' αυτό δεν θα πρέπει στα κριτήρια που θα χρησιμοποιήσουμε για να αποφασίσουμε αν θα πετύχει όχι, ή αν επέτυχε μάλλον ή όχι η Κοπεχάγη, δεν θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ακριβώς και τις δεσμεύσει και τις προσπάθειες που θα πρέπει να κάνουν η Κίνα, η Βραζιλία και η Ινδία. Merci beaucoup, Edith Estrella. Ευχαριστώ κυρία Στρέλα. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στη μορφή χρηματοδότησης που θεωρώ ότι είναι ακόμα πολύ αόριστη και ακαθόριστη, ενώ είναι ένα κρίσιμο ζήτημα ώστε να καταφέρουμε να πετύχουμε την ε, σφαιρική συμφωνία τα κονδύλια είναι ψηλά, αλλά δεν είναι συνενετικά αυτά που ακούμε. Ορισμένοι μιλάνε για 100 εκατομμύρια, άλλοι μιλάνε για 15, για 15 δις το χρόνο. Ε, και άρα λοιπόν, πότε, πόσα θα χρειαστούν για να στηρίξουμε την προσαρμογή στις αναπτυσσόμενες χώρες. Και έπειτα, ποιος θα τα χρηματοδοτήσει όλα αυτά, διότι προφανώ δεν μπορεί να είναι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ε, τρίτον, πέρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλα αυτά θα έρθουν ε, από την αναπτυξιακή βοήθεια που ήδη είναι προγραμματισμένη θα υπάρξουν παραπάνω κονδύλια. Ο κύριος Πρόντι. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε. Εσείς γνωρίζετε ποια είναι η θέση μου σε σχέση με την έλλειψη μιας ε, ρήτρα ισότητας στην πρόταση για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Ε, στις ε, διαπραγματεύσει τη Βαρκελόνη, ορισμένες αφρικανικές χώρες βγήκαν από τη συζήτηση. Τι σχόλιο μπορείτε να κάνετε, Επίτροπε, από αυτού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Κορίν Λεπάζ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Το ερώτημά μου αφορά την διαρροή άνθρακα. Θέλω να ξέρω αν θεσπίζοντας τον κατάλογο η Κομισιόν έχει μια ιδέα ή αν είχε κάνει κάποιες ε, προεκβολές για να προσπαθήσει να δει ακριβώ ε, τι αντιπροσωπεύει κάτι τέτοιο και αν έχει κάποια συγκεκριμένη ιδέα για τον αριθμό των τόνων άνθρακα που θα διέφευγε από το σύστημα πληστηριασμών και ποιες θα ήταν οι πραγματικές συνέπειες αυτού του καταλόγου. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, παρακολουθούμε το έργο του Επιτρόπου του κυρίου Δήμα και ευχόμαστε την ανανέωση της θητείας του. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε μια διαρκή προσπάθεια να υποβαθμιστεί η νομική δέσμευση που θα απορρέει από το COP15, καθώς στην αρχή μιλάγαμε για συνθήκη, τρίτη, μετά για πλαίσιο, framework και τώρα για μια απλή πολιτική δέσμευση declaration, όπως είπε χθε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Βαρκελόνη. Το κρίσιμο ζήτημα σχετικά με τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν ώψη της συνδιάσκεψης της Κοπεχάγης είναι από ό,τι φαίνεται η απροθυμία της να υιοθετήσει τις προτάσεις της επιστημονικής κοινότητας και να επιδείξει έναν ηγετικό ρόλο στην παγκόσμια προσπάθεια ενάντια στην κλιματική αλλαγή. Η επιστημονική ομοφωνία αποτυπώνεται στην έκθεση του IPCC ε, ότι οι αναπτυγμένες χώρες θα πρέπει να μειώσουν τις εκπομπές τους μέχρι και 40% το 2020 σε σχέση με το 1990 και 80% μέχρι το 2050 αν είναι να καταπολεμήσουμε ε, αποτελεσματικά τις κλιματικές αλλαγές. Ε, επίσης, ε, σε περίπτωση επίτευξης ε, ε, διεθνούς συμφωνίες, οπότε και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ανεβάσει το στόχο μείωση σε 30% και πλέον. Ε, ρωτώ, ποιες είναι εκείνες οι πολιτικές και τα μέτρα που η Επιτροπή θα πρότεινε να αναθεωρηθούν. Για ποιο λόγο η Επιτροπή αντιτίθεται σε δεσμευτικούς στόχους ενεργειακής αποδοτικότητας και τέλος αν έχει συζητήσει ε, η Επιτροπή το θέμα αυτό με τις εθνικές κυβερνήσεις και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Η κυρία Χουμνέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Επανειλημμένα σήμερα είπαμε ότι ο κατάλογος αυτός ε, θα αναθεωρηθεί μετά την Κοπενχάγη. Ακούσαμε επίσης ότι έχουμε στόχο μείωσης 20%. Ε, πώς θα τον αναθεωρήσουμε τον κατάλογο μετά την Κοπενχάγη. Θα στεθούν κάποιοι κλάδοι ή θα αφαιρεθούν άλλοι που είναι ήδη στο κατάλογο. Προς ποια κατεύθυνση θα πάει η αναθεώρηση. Γιατί μας είπαν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα φέρει νέο κατάλογο μετά τη διάσκεψη. Και από εκεί και πέρα έχουμε ένα σχέδιο εναλλακτικό. Αν οι περισσότεροι ας πούμε συμμετέχοντες δεν δεχτούν τις προτάσεις μας. Τι θα κάνουμε. Θα επαναξεταστεί ο κατάλογος και προς ποια κατεύθυνση. Ευχαριστώ. να Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Καταρχήν, όσον αφορά τη χρηματοδότηση, μιλάμε για δύο περιόδους, 2010 με 2012 και τη δεύτερη που ξεκινάει από το 2013. Κύριε Επίτροπε, συμφωνείτε με την ιδέα ότι στην πρώτη περίοδο 2010-2012 τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα πρέπει να συμβάλλουν στη χρηματοδότηση σε, χρημα... εθελοντική βάση και σε τι βαθμό η Επιτροπή, κατά πόσο η Επιτροπή συμφωνεί μετά το 2013 με βάση την ε, οικονομική δύναμη των διαφόρων κρατών μελών να εκπονηθεί κλίδα κατανομής ε, του κοινού φόρτου. Τρίτη ερώτηση. Όσον αφορά το διάστημα μέχρι το 2012 και τις ποσοστώσεις ε, που ήδη έχουν πολιθεί για μετά το 2013, ο Επίτροπος συμφωνεί με τη μέθοδο αυτή και τέλος, το 1987 καθορίστηκε 8% μείωση των ε, εκπομπών. Ε, κυρία Ντεμπρούν, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο που ήρθε και ε, για τα καλά του λόγια επίσης για το ψήφισμα που προτείνουμε για το ΚΑΠ15. Ε, θέλω να σας ρωτήσω κάτι ειδικά για το ψήφισμα. Πώς βλέπετε την παράγραφο 18 που μιλά για τη συλλογική συνεισφορά προς τις ανάγκες των τρίτων χωρών που δεν θα πρέπει να κάνω από 30 δισεκατομμύρια μέχρι το 2020. Και μετά ποια είναι η θέση που θα πρέπει να λάβουμε για το πρωτόκολλο του Κιώτο και τη διάδοχη ε, κατάσταση. Και σε σχέση με τα σχόλια και τα όσα συζητήθηκαν στην Μπαγκόκ. Οπότε φαίνεται ε, εκεί ε, μάλλον προωθείται μια ενιαία και συνολική συμφωνία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αναρωτιέμαι αν μπορείτε να εξηγήσετε ποια ακριβώς στοιχεία χρησιμοποίησε η Επιτροπή κατά την αξιολόγηση των ε, στόχων της Νορβηγίας, Ισλανδίας και Ελβετίας. ποια ήταν τα δεδομένα και ποια ήταν η πηγή τους. Και επίσης, τι δεδομένα χρειάζεστε ακόμα για να κάνετε την ίδια αξιολόγηση για την Βραζιλία, την Αυστραλία, τη Ιαπωνία, χώρες δηλαδή που επίσης έχουν στόχους μείωσης. Και είμαι βέβαιος ότι παρότι δεν έχετε τα δεδομένα αυτά ακόμα, θα έχετε κάποια ε, ένδειξη σχετικά με το προς ποια κατεύθυνση πηγαίνουμε. Μπορείτε να μας πείτε αν κάτι τέτοιο θα οδηγήσει σε ε, μικρότερο ή μεγαλύτερο κατάλογο για την ε, μετακατάσταση των εκπομπών. Και Επίσης, αναφερθήκατε στον στόχο των 2 βαθμών Κελσίου. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι, αναπτυσσόμενες χώρες, όλες οι αναπτυγμένες χώρες ε, θα πρέπει να ε, μειώσουν εκπομπές σε 20 40%. Αυτό τι σημαίνει για τις ΗΠΑ. Παραμένει ο στόχος αυτός ρεαλιστικός. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ ο Καρλ Σλίτερ. Καταρχήν ε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για μια πενταετία καλή συνεργασία και πολύ υγιών συγκρούσεων. Πρώτη μου ερώτηση, πώς ε, μπορούμε να αποφύγουμε οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, να αποδυναμώσουν τη συμφωνία και η ε, γερουσία τους να την καταψηφίσει. Δεύτερον, πιστεύετε ότι με 20% μείωση στην Ευρώπη μπορούμε να πετύχουμε το στόχο των 2 βαθμών Κελσίου δεν πρέπει ούτως ή άλλως να προχωρήσουμε πέρα από το 20% και ποια είναι τα κριτήρια για το 30% διεθνής αν έχουμε διεθνή συμφωνία όπου οι Ηνωμένε Πολιτείε και άλλοι να μην συμμετέχουν, πάλι θα επιδιώξουμε το 30%. Και όσον αφορά τη μετακατάσταση των εκπομπών, πώ θα αναθεωρήσετε τον κατάλογο όταν συμμετάσχουν και άλλες χώρες. και πώς μπορείτε να αποφύγετε να μην ε, ξαναεπενδύουν οι επιχειρήσεις. Ε, δεν θα ήταν καλύτερο να έχουμε ένα κατάλογο που να βασίζεται στους 10 καλύτερους και τι θα κάνετε σε περίπτωση που ένας ε, τομέας έχει έναν παραγωγό ή έναν υποτομέα μέσα ε, στα πλαίσια ενός τομέα. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν έχουμε ένα λείπασμα που δεν ε, πληρεί τα κριτήρια, ε, θα θεωρείται ότι το σύνολο του τομέα μπορεί να αποτελεί σε αντικείμενο μετακατάσταση των εκπομπών. Κύριο Σκυλακάκη, παρακαλώ. Κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ επίσης και σαν την χρέωση να πω ότι η χώρα μας αισθάνεται υπερήφανη για τη δουλειά που έχετε κάνει αυτά τα τελευταία χρόνια. Θα πω όμως ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα. Στην τελευταία διάσκεψη των G20 η, ελήφθη η απόφαση να ξεκινήσει η περικοπή των επιδοτήσεων στα καύσιμα που δίνονται από μία σειρά χωρών. Το θέμα αυτό είναι τεράστιο. Μιλάμε για 330 δισεκατομμύρια ε, δολάρια το χρόνο επιδοτήσεις, τάξη μεγέθους. Η κατάρρηση δε αυτών των επιδοτήσεων κατά τον ΟΣΑ και την International Energy Agency μπορεί να οδηγήσει σε κατά 10% περιορισμό των παγκόσμιων εκπομπών μέχρι το 2050. Τώρα, πού πηγαίνουν αυτές οι επιδοτήσεις. Μιλάμε κυρίως για κατανάλωση, επιδότηση κατανάλωση βενζίνης, μεσαίων στρωμάτων, χωρών πετρελαιοπαραγωγών και αν θυμηθείτε τα μποτιλιαρίσματα που υπάρχουν στις μεγάλες μητροπόλεις, είναι ακριβώς εκεί. Το ερώτημα λοιπόν είναι αυτή η από πλευράς ενεργειακής απόδοσης ακραία ε, σπατάλη θα τεθεί στην Κοπενχάγη ως ισχυρή κατεύθυνση στα προγράμματα τα εθνικά ή θα την αφήσουμε ανέγγιχτη. Ευχαριστώ κύριε Κλάς. Ευχαριστώ. Κύριε Επιτροπέ η Κοπενχάγη δεν θα είναι απλή υπόθεση, διότι, και αυτό είναι πεποίθηση του Κοινοβουλίου, χρειαζόμαστε όλους το πλευρό μας. Τι θα γίνει με τα χρήματα που διατίθενται στις αναπτυσσόμενες χώρες και που θα αυξηθούν. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σωστά μεταφορά τεχνογνωσίας, σχέδια υπέρ του περιβάλλοντος από πλευράς των κρατών αυτών. Θα πρέπει όμως νωρίτερα να ξεκινήσουμε από την παιδεία, από τη συνειδητοποίηση των πληθυσμών, για να είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα επαναληφθούν τα σφάλματα που κάναμε εμείς και που θέλουμε εμείς να διορθώσουμε ως στρεβλά. Στην Πουρκίνα Φάσο, ας πούμε, θέλει κάθε σπίτι να ε, έχει ε, μία αιστεία, ε, ένα τζάκι. Καλό είναι αυτό, αλλά μήπως πρέπει να σκεφτούμε και την ηλιακή ενέργεια. δηλαδή να βοηθούν οι ανεπτυγμένες χώρες, οι αναπτυσσόμενες, αλλά ακόμα δεν έχουμε καταλήξει σε αυτό. Δεν υπάρχει συνειδητοποίηση ότι είμαστε όλοι στην ίδια μοίρα ότι και θα πρέπει και εμείς να βοηθήσουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα περιστώ σε μία ερώτηση. Είχα τρεις για τη μετεκατάσταση εκπομπών που πρέπει να ψηφίσουμε σε λίγο για τη λίστα. Είναι σημαντικό στην Ευρώπη να λαμβάνουμε υπόψη τους τομεί που θα πληγούν πάρα πολύ αν δεν υπάρξει συμφωνία. Βεβαίως όλοι ελπίζουμε σε συμφωνία. Είπε ο Επίτροπος ότι θα ε, προσαρμοστεί ο κατάλογο και παρέπεμψε στο συμπέρασμα 22 του Συμβουλίου, αλλά δεν λέει ημερομηνία εκεί. Αν κοιτάξει κανεί το κείμενο, της νομοθεσίας γίνεται λόγος για τον Ιούνιο του 2010. Είπε επίσης ο κύριος Επίτροπος ότι θα γίνει αυτό σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο. Άρα συναπόφαση. Αυτό μπορεί να χρειαστεί και να διαρκέσει και 1,5 και 2 χρόνια. Κύριε Επίτροπε, πώς βλέπετε το χρονοδιάγραμμα, πώς το φαντάζεστε, αν φτάσει μόλις τον ε, Ιούνιο η πρόταση, χαιρετίσματα, θα πάει πολύ χρόνο. Κύριε Ρόσπα. Θα ήθελα να επανέλθω στην χρηματοδότηση. Κύριε Δήμα, λέτε ότι οι ανεπτυγμένες οικονομίες ε, θα πρέπει να, αποτελέσουν, να παίξουν σημαντικό ρόλο όσον αφορά την ε, μείωση των εκπομπών. Εσείς ποιες οικονομίες έχετε κατά νου. Δεύτερον, η Κομισιόν έχει αρχίσει να εφαρμόζει παρόμοιους στόχους για το πόσιμο νερό, ε, όπως και για την ποιότητα του αέρα. Ευχαριστώ. Κατρίν Σουγιέ. Madame Sui. Oui, merci, Président. Très vite. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ σύντομα ε, ναι, περικόπουμε τις εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα, αλλά θα πρέπει να διατηρήσουμε τους ωκεανούς και τα δάση που είναι τα φυσικά, οι φυσικοί πόροι ε, της γης. Αναφέρθηκε η αποδάσωση, εμείς ε, τιμωρούμαστε διπλά. Ε, Καίγονται τα δόντια, τα δάση, τα δάση, μάλλον η φωτιά εκπέμπει διοξίδιο του άνθρακα. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν να έχουμε θετικά αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε που έχετε σφαιρική εικόνα του προβλήματος, δηλαδή από μια πλευρά εκπομπή και από την άλλη συντήρηση όλων των φυσικών ζωνών που επιτρέπουν να απορροφάτε το διοξίδιο του άνθρακα. Ουφ, 27 μιλήσατε. Ευχαριστώ και τους 28 ε, για την πειθαρχία. Πολλές ερωτήσεις, καλές σημαντικές, δεν ξέρω πώς θα καταφέρετε να τις απαντήσετε. Ε, σημειώσατε, βλέπω, όλες τις ερωτήσεις και όλους τους ερωτώντες. Ελπίζω να ε, απαντήσετε σε σύνοψη. Ίσως το πρώτο αυτό το θέμα για τη λίστα της μετεκατάστασης εκπομπών Carbon Leakage, γιατί θα ψηφίσουμε σε λίγο γι' αυτό. Και όσα μπορείτε από τα υπόλοιπα, νομίζω ότι θα Πρέπει να ζητήσουμε από τους διερμηνείς λίγα λεπτά να παραμείνουν για την ψηφοφορία μετά τις 12.30. Εγώ υποτίμησα ε, το ρολόι εδώ, το, το, επίσημο που πάει πέντε λεπτά πίσω. Εν Κύριε Πίτροπε, έχετε το λόγο. On ε, carbon leakage, ε, don't Για τη διαρροή άνθρακα. Μην ξεχνάτε ότι αυτό που εφαρμόζουμε εδώ είναι αυτό που συμφωνήθηκε στην διαδικασία συναπόφασης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από το Συμβούλιο. Διότι η αρχική μας πρόταση δεν ήταν ακριβώς αυτή που έχουμε σήμερα. Ωστόσο, καθώς εφαρμόζουμε τώρα αυτή την οδηγία, θα ήθελα να δηλώσω ότι είμαστε πολύ, προσέχουμε πάρα πολύ ώστε να ακολουθήσουμε τα όσα μας λένε οι νομικοί μας σύμβουλοι. Και Να είμαστε σύμφωνοι με τα όσα μας λένε οι νομικές μας υπηρεσίες και καταλαβαίνω πως και εσείς ζητήσατε νομική συμβουλή για τα θέματα αυτά. Δεν την ε, έχω δει ε, τα απορίσματα της Ευρωπαϊκής σα Επιτροπής αλλά, ε, του νομικού, των νομικών συμβούλων, αλλά φαντάζομαι ότι είναι παρόμοια με αυτά που εμείς προτείνουμε. Το βασικό θέμα είναι αν μπορεί αυτός ο κατάλογος να αναθεωρηθεί ή όχι, αν μπορούν να προσθεθούν κάποιοι τομείς ή να αφαιρεθούν. Και τα δύο μπορούν να συμβούν μπορούν να γίνουν σύμφωνα με την αξιολόγηση που θα γίνει το Ιούνιο του 2010 μετά από την αξιολόγηση της Συμφωνίας της Κοπεχάγης και βέβαια ανάλογα με τα αποτελέσματα αυτής της συμφωνίας και βεβαίως μέσω της διαδικασίας συναπόφασης. Αυτό είναι που αποφασίστηκε όταν συζητήσαμε την οδηγία και αυτό οφείλουμε να κάνουμε. Αυτή είναι λοιπόν η απάντησή μου και ελπίζω πως θα ψηφίσετε σύμφωνα με αυτό που πιστεύετε ότι είναι το πιο σημαντικό ώστε να μην διακοπεί η διαδικασία. Άκουσα ερωτήσεις αλλά και δηλώσεις πολλές που ήταν ενδιαφέρουσες. Θα προσπαθήσω να τις ομαδοποιήσω όσο μπορώ. Ξεκινώ, για παράδειγμα, με το ερώτημα που μου έθεσε ο Βιτόριο Πρόντι σχετικά με τη χθεσινή άρνηση των Αφρικανικών χωρών να συνεχίσουν τη συζήτηση στην Βαρκελόνη. Μέσα στο πλαίσιο της, των διαπραγματεύσεων για το Κιώτο, πριν οι αναπτυσσόμενες χώρες δεσμευτούν για αριθμούς, για στόχους. Και ναι, βεβαίω θα πρέπει να πω ότι συμφωνούμε απόλυτα με τι αφρικανικέ χώρε και εμεί αυτό επιθυμούμε. Αλλά το να πάμε στο άλλο άκρο και να διακόψουμε τις συζητήσεις που αφορούν και άλλα σημαντικά θέματα, δεν νομίζω πως είναι ο ιδανικός τρόπος πρόθεσης της συζήτησης. Και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο ε, σε αυτήν την αφρικανική ομάδα ο βασικός ρόλος το βασικό ρόλο έπαιξαν όχι μόνο αφρικανικές χώρες όπως το Σουδάν, αλλά και η Σουδική Αραβία, η Βολιβία, η Βενεζουέλα, χώρες που δεν ε, παίζουν πραγματικά επικοδομητικό ρόλο στι διαπραγματεύσει. Αλλά ελπίζω πως αυτό θα ξεπεραστεί. Η μία σχετική ερώτηση αφορούσε την παράπονα ορισμένων χωρών στην Πανκόγκο, ιδιαίτερα την Ινδία, πως οι αναπτυσσικμένες χώρες σκοτώνουν το Κιώτο. Αυτό δεν είναι ασύμβατο με αυτό που λέμε, ότι προτιμούμε ένα εννέο νομικό κείμενο και σας το εξήγησε. Το προτιμούμε, είπα, δεν λέμε ότι το αποκλείουμε οτιδήποτε άλλο. Αλλά το να σκοτώσει κανείς το Κιώτο δεν σημαίνει, το ότι σκοτώνουμε το Κιώτο δεν σημαίνει ότι είναι κατηγορία κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί είμαστε οι πιο στεναροί υποστηρικτέ του. Ξέρετε πόσο πολύ έχουμε δουλέψει και ανοίγω και μια παρένθεση και σας ευχαριστώ για την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε κατά τη διάρκεια αυτών των ετών και τα όσα που καταφέραμε στις κλιματικές αλλαγές αλλά και σε άλλα περιβαλλοντικά ζητήματα επετεύθη με τη δική σας ενεργή υποστήριξη. Χωρίς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την υποστήριξη των ΜΚΟ δεν θα είχαμε καταφέρει τα αποτελέσματα που έχουμε. Μάλιστα και αυτό που είπε ο πρόεδρος Μπαρόζο, ότι μεγαλύτερη το μεγαλύτερο κληροδότημα ε, μακράν είναι αυτό που πετύχαμε με για τις κλιματικές αλλαγές σε αυτή τη θητεία της Κομισιόν, πραγματικά ήταν πολύ σπουδαίο. Θα παρακολουθώ πάντα τι θα γίνει στο μέλλον, και, γιατί το κλίμα θα κυριαρχήσει όχι μόνο στις ζητήσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και διεθνώς, όχι λόγω για περιβαλλοντικούς λόγους αλλά και για οικονομικούς λόγους και για λόγους ασφαλείας και για, άλλα, ένα, και για έναν άλλο σωρό λόγων όπως η υγεία για παράδειγμα. Και είμαι βέβαιος πως η Κομισιόν θα συνεχίσει στην ίδια γραμμή. Στον ε, φίλο μου Τρεμόπουλο από την Ελλάδα όσον αφορά το ότι η δική μου εντολή θα ανανεωθεί. Ξέρετε πως είχαμε εκλογέ τελευταία. Οι κυβερνήσεις ε, αποφασίζουν όχι με βάση την απόδοση του καθενός, αλλά με βάση την πολιτική του θέση. Εκεί είμαι βέβαιο ωστόσο, ότι η ελληνική κυβέρνηση θα επιλέξει έναν καλό επίτροπο που θα μπορέσει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων ε, σε οποιοδήποτε χαρτοφυλάκιο για να αναλάβει. Τώρα, για το κλίμα και το Κιώτο. Όπως σας είπα, το Ευρωπαϊκή Ένωση είναι βασικός υποστηριχτής του Κιώτο και πολύ στεναρό μάλιστα. Ενεργά έχουμε υπερασπίσει την επικύρωση του Κιώτο. Και είχαμε το πρωτόκολλο του Κιώτο από το Φεβρουάριο του 2005 που εφαρμόστηκε, του 16 Φεβρουαρίου 2005. Και αυτό χάρη στις διαπραγματεύσεις που κάναμε, την πίεση που, και την πειθό που, ε, με την οποία ενεργήσαμε κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ετών. Στη συνέχεια, εφαρμόζουμε το Κιώτο. Έχουμε το σύστημα εμπορίας των εκπομπών που λειτουργεί και λειτουργεί με επιτυχία. Και έχουμε επίσης επενδύσεις σε μηχανισμούς καθαρής ενέργειας που είναι ακόμα ένας μηχανισμός για την αγορά άνθρακα και επενδύουμε σε ολόκληρο τον κόσμο και έχουμε επενδύσει περίπου 80% όλων των προγραμμάτων και καθαρών μηχανισμών από την Ευρωπαϊκή Ένωση προέρχονται πράγμα που με τη σειρά του χρηματοδοτεί το Ταμείο της Προσαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών που με τη σειρά του στηρίζει προγράμματα προσαρμογής στις αναπτυσσόμενες χώρες. Το 70% των χρημάτων εκεί προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επίσης έχουμε οικοδομήσει τη μελλοντική μας νομοθεσία μάλλον την νομοθεσία μας για το μέλλον μέχρι το 2020, το πακέτο κλίματος και ενέργειας στην αρχιτεκτονική του Κιώτο και στις ιδέες του Κιώτο. Άρα λοιπόν υποστηρίζουμε το Κιώτο και στο μέλλον στο μέλλον, στη μελλοντική συμφωνία της Κοπεχάγης, έχουμε σαφώς δηλώσει πως επιθυμούμε αυτή να βασιστεί στο Κιώτο και η βασική αρχιτεκτονική και μηχανισμοί του Κιώτο να μεταγραφούν και στην επόμενη μελλοντική συμφωνία της Κοπεχάγης. Ένα μόνο δεσμευτικό κείμενο, γιατί κάποιος, ε, νομίζω ο Κρις Ντέιβις στην αρχή με ρώτησε για την πολιτική συμφωνία και θα, το, θα έρθω σε αυτό, ένα ενιαίο κείμενο θα είναι καλύτερο για λόγους συμμετοχής, διότι ένα ενιαίο κείμενο θα επικυρωθεί ταυτόχρονα, ενώ αν έχουμε δύο-τρία έγγραφα η διαδικασία επικύρωσης ε, ίσως να είναι ε, διαφορετική και δεν θα έχουμε ίσως τη συμμετοχή όλων των χωρών ταυτόχρονα. Συνοχή, συνέπεια, να έχουμε ένα έγγραφο, δεν θα υπάρχουν ε, λόγοι για ασυνέπεια ανάμεσα στις παρόμοιες νομικές διατάξεις Αυτό είναι όμως βασικά, εντάξει θα συντομεύσω, αλλά είναι βασικά πράγματα. Είναι η βάση της συζήτησή μας τώρα, αν θέλουμε, αν χρειαζόμαστε ένα ενιαίο δεσμευτικό κείμενο ή όχι, αν θα έχουμε τροποποίηση του Κιώτου, πράγμα που είναι απαράδεκτο για τους Αμερικανούς π.χ. Και, για το, και κατά πόσο οι χώρες θα συμμετέχουν οι αναπτυγμένε και αναπτυσσόμενε με διαφοροποίηση τη ουσία όσον αφορά τι δεσμεύσει, αλλά όχι ε, τη νομική μορφή. Και αυτή είναι η βασική μα διαπραγματευτική διαφορά. Λοιπόν, αυτό που χρειαζόμαστε είναι ένα κείμενο ενιαίο και δεσμευτικό. Αλλά δεν αποκλείουμε, αν επιμείνουν άλλοι εθνεί εταίροι, να έχουμε δύο παράλληλα κείμενα, σχεδόν ταυτόσημα, για να αποφύγουμε να βαφτιστεί το νέο κείμενο και το ναι και το όχι. Ξέρετε ότι αυτά τα πράγματα είναι πολύ σημαντικά στι Ηνωμένε Δεν θέλουν να ακούσουν λέξη για το Κιώτο, ούτε το συζητούν, ούτε τίποτα δεν σηκώνουν για το Κιώτο. Τώρα, εάν θα έχουμε πολιτική συμφωνία αν θα την επιδιώξουμε. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα συμπεράσματά του, αλλά και το Συμβούλιο Υπουργών ε, περιβάλλοντος στα συμπεράσματά του στις 21 Οκτωβρίου μιλούν για ε, φιλόδοξη παγκόσμια συνολική δεσμευτική συμφωνία. Παγκόσμια σημαίνει όλες τις χώρες του κόσμου. Αναπτυγμένες, αναπτυσσόμενες, ανάλογα με το πώς γίνεται αυτή η διάκριση των αρμοδιοτήτων συνολικό πλήρες που σημαίνει όλου του κλάδους και τη δασοκομεία και τις θαλάσσιε μεταφορές και τις αερομεταφορές που δεν είχαν καλυφθεί από την προηγούμενη διεθνή συμφωνία ή τι συμφωνίες και παρένθεση. Κατά τα άλλα εμείς είμαστε και πάλι οι πρώτοι στον κόσμο που έχουμε στόχο 10% για την ε, αεροπορική βιομηχανία και 20% για τις θαλάσσιες μεταφορές και συζητήθηκε και στο Συμβούλιο Περιβάλλοντος και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Έτσι λοιπόν θέλουμε παγκόσμια, συνολική, πλήρη, ε, φιλόδοξη συμφωνία. Φιλόδοξη τι σημαίνει. Το στόχο του κάτω των δύο βαθμών Κελσίου που συμφώνησαν ηγέτες των ε, μεγάλων οικονομιών ε, του κόσμου στη Λάκουιλά της Ιταλίας τον Ιούλιο. Είπα Κίνα, Ινδία, βεβαίως Ευρωπαϊκή Ένωση, τα έχουν συμφωνήσει αυτά. Είπαμε, σύμφωνα με την επιστήμη, εάν δεχτούμε δύο βαθμούς Κελσίου, αλλιώς θα έχουμε ανεπανόρθωτες ε, και ολέθριες επιπτώσεις. Άρα θα πρέπει να περιορίσουμε την αύξηση της θερμοκρασίας μέχρι το 2050 στους δύο βαθμούς σε σχέση με ε, θερμοκρασίες πριν ε, τις βιομηχανικές εποχές. Αυτά τα έχουμε και στο Συμβούλιο λοιπόν ε, ως συμπεράσματα και είναι η διαπραγματευτική θέση της Ένωσης για την Κοπεχάγη. Αυτά επιδιώκουμε. Τώρα, ως προς την πολιτική συμφωνία. Θα διαβάσατε στις εφημερίδες σήμερα ή εχθές ότι ο Δανός Πρωθυπουργός όχι ως Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ως πρόεδρος της COP15 της Κοπεχάγης, έχει πει ότι πάλι θέλουμε φιλόδοξη, πολιτικά, δεσμευτική συμφωνία πλέον, που να συμπεριλαμβάνει ε, τους βασικούς μεγάλους συνασπισμούς, ας πούμε, με τα μπλοκ και τις δέσμες ε, που χρειάζεται για να φτάσουμε σε αυτό το στόχο κάτω των 2 βαθμών Κελσίου. Αυτό είναι κάτι που είπε ο Δανός λοιπόν Πρωθυπουργό. Δική του εκτίμηση είναι. Εμείς αγωνιζόμαστε για ε, νομικά δεσμευτική συμφωνία, όχι πολιτικά. Λυπάμαι, αλλά έχω τόσες πολλές ερωτήσεις και θα ήθελα να απαντήσω στις περισσότερες, αλλά τι να κάνουμε. Δεν το επιτρέπει ο χρόνος. Το γνωρίζω. Σας ευχαριστώ και πάλι πολύ. Ε, σας ευχαριστώ για την εξαιρετική συνεργασία και είμαι βέβαιος ότι όλα αυτά που επιτύχαμε όλα αυτά τα χρόνια μαζί θα είναι πολύ σημαντικά για το πλανήτη μας και για την Ευρώπη και παρακαλώ ας μην λησμονούμε και τελειώνουμε αυτό. Κάτι που είπε ένας, μάλλον ένας Ιταλός συνάδελφος μου είπε κάτι, ότι δεν νοιαζόμαστε για τη βιομηχανία μας. Το αντίθετο, και τη νοιαζόμαστε και τη φροντίζουμε και την πονάμε. Γι' αυτό φτιάξαμε και αυτό τον κατάλογο με την κατάσταση εκπομπών για carbon leakage. Και επίση όχι μόνο αυτό, έχουμε βάλει και στο ETS μια πρόβλεψη που προβλέπει και άλλα μέτρα ακριβώ. Σε περίπτωση που δεν καταλήξουμε σε διεθνή συμφωνία και έχουμε προβλήματα ανταγωνιστικότητας στο μέλλον. Άρα είναι θέμα εκτίμησης της Συμφωνίας Κοπεχάγη για να δούμε τι θα συμφωνηθεί από εκεί και πέρα σε λεπτομέρειες και άλλο σημαντικό θέμα είναι ότι το πακέτο για την ενέργεια και το κλίμα που έχουμε είναι πολύ σημαντικό για την ευρωπαϊκή οικονομία, για την ευρωπαϊκή βιομηχανία και ανταγωνιστικότητα, γιατί δίνει κίνητρα για επενδύσεις, για οικοκαινοτομία και μην ξεχνούμε ότι στην ευρωπαϊκή οικονομία η λεγόμενη πράσινοι τομεί είναι εκείνοι που αναπτύσσονται με ταχύτερου ρυθμούς και δημιουργούμε πολλές πράσινες θέσεις απασχόλησης. Και αυτό έχει γίνει και μόδα παγκόσμια. Ξαφνικά και ο Ομπάμα πρασίνησε. Έχει τα πράσινα σχέδια ανάπτυξης, η Κίνα, το ίδιο η Νότια Κορέα επίσης. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό να είμαστε πιο φιλόδοξοι και είμαστε. Αλλά το 70% του σχεδίου ανάκαμψης η Νότια Κορέα το επενδύει στις πράσινες τεχνολογίες. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ κύριε Δήμα. Κύριε Επίτροπε, δεν ξέρω αν είναι η τελευταία φορά που έρχεσαι στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Πρέπει να σας ευχαριστήσω εξ ονόματος. Θα τα πούμε στην Κοπεχάγη. Εντάξει, εντάξει εκτός αν μέχρι τότε ε, θα έχει αναλάβει η Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, Α, νόμιζα θα μου λέγατε, θα παραμείνω επίτροπο στην Κοπεχάγη, μέχρι την Κοπεχάγη. Πιστεύω ότι 1η Δεκεμβρίου θα τεθεί σε ισχύ η συνθήκη, αλλά από ό,τι φαίνεται μέχρι να γίνουν όλες οι ακροάσεις 1η Ιανουαρίου θα αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βεβαίως βεβαιω ραντεβου στην Κοπεχάγη και με χαρά να σας δούμε εκεί γιατί είστε πραγματικά προσιλωμένο και στρατευμένο σε αυτά τα θέματα του περιβάλλοντο και ιδιαίτερα τη προστασία από την κλιματική αλλαγή. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε εδώ και για τη συνεργασία σα την τελευταία πενταετία με το Κοινοβούλιο. Και καλή δύναμη και ό,τι επιθυμείτε. Äh, λοιπόν, Πέντε λεπτά ακριβώς διάλειμμα με το ρολόι και μετά ψηφίζουμε. now. Για τα βρώνει πολιτικές ομάδες. Yeah. Five minutes, the clock is uh, running. Λοιπόν, πέντε λεπτά με το ρολόι, το έχω βάλει. So, kollegen, Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, πέρασαν τα πέντε λεπτά και ερχόμαστε στην ψηφοφορία. Επειδή είναι πολύ σημαντικό, θα πρέπει να κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία για να δούμε ποιοι και μάλλον πόσοι ψηφίζουν από κάθε πολιτική ομάδα. Ε, δοκιμαστική ψηφοφορία και πάλι να δούμε αν θα έχει ήλιο τα Χριστούγεννα. Ναι, όχι, εποχές αν θα έχουμε ηλιόλου στα Χριστούγεννα. Λοιπόν, πριν βγει ο ήλιος στα Χριστούγεννα, το ΕΛΚ περσεύουν πέντε από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Να πει ο συντονιστή ποιο θα ψηφίσει και ποιο δεν θα ψηφίσει. Ένα. Βρείτε πέντε να του διώξετε. Και οι σοσιαλιστέ, ένα περσεύει. Εντάξει. Το ΕΛΚ ακόμα δύο παραπάνω και από τους σοσιαλιστές ένας παραπάνω. PPE, fine. Τώρα είναι εντάξει το ΕΛΚ αριθμητικά. 61 μέλη έχουμε που δικαιούνται να ψηφίσουν. Λοιπόν, δοκιμαστικά ψηφίζουμε, θα έχει ήλιο τα Χριστούγεννα. Τώρα. Πάμε στην κανονική ψηφοφορία που αρχίζει τώρα, η επίσημη. We have still EPP and... ΕΛΚ και οι σοσιαλιστές έχετε ένα παραπάνω. S&D one too much. S&D ένας παραπάνω. Πού λέει η κυρία Μακάβα. 16, yeah. 16 είμαστε. machine says one too much. machine says one too much. That's one. The machines That's one too much. Yes, now it's fine. Yeah. Now it's fine. Τώρα είναι εντάξει, γιατί είχατε κάρτα στο μηχάνημα, ακόμα και αν δεν ψηφίζατε. Πέρας. Αποτέλεσμα. 19 υπέρ, 39 κατά και μία αποχή. Άρα το ψήφισμα απορρίπτεται από την Επιτροπή. Καλώς, ευχαριστώ πολύ. Μεσημεριανό διάλειμμα, συνέχεια στις 3.